Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας. Άστο. Find Παρακαλώ καθίστε. Και ετοιμαστείτε και θα μιλήσω σου ειδικά. Εάν δεν καταλαβαίνετε λοιπόν τα σου ειδικά, Μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά σας. Oh, that really silenced the audience. I mean. Ξαφνικά σοπάσατε όλοι. Θα το λέω πιο συχνά. Γιατί όλοι τότε θα σοπαίνουν. Καλώ ήρθατε στη συνεδρίασή μα. Είναι μια συνεδρίαση με μεγάλο ενδιαφέρον, η σημερινή. Πρόκειται για ένα σεμινάριο για τη συμμετοχή των γυναικών στις ανώτατες ε, διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες συσυγμένες στο χρηματιστήριο. Χαίρομαι που έχουμε ένα μακρύ κατάλογο μιλητών που θα παρουσιάσουν ε, τις απόψεις τους που φαντάζομαι θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Είσαστε τόσοι πολλοί που θέλετε να μιλήσετε που δεν πρέπει να μιλήσω πολύ. Έχουμε τους εισηγητές καταρχήν που πρέπει να πάρουν το λόγο προφανώς και συνεχεία Έχουμε και τους ε, προσκεκλημένους ομιλητές. έχουμε και εκπρόσωπο, την, ε, εκπρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Θέλω να καλωσορίσω θερμά όλους τους ομιλητές. Και πριν περάσουμε στο πρώτο πάνελ, να σας υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να σεβαστείτε το χρόνο, γιατί υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μιλήσουν. Κάθε ομιλητή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα πέντε λεπτά. Ξεκινάμε την κυρία Κράτσα Τσαγκαροπούλη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Θεωρώ και εγώ ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σήμερα η συνάντηση αυτή που έχουμε και το πρόγραμμα όπως έχει προετοιμαστεί και χαίρομαι πολύ που καταφέραμε να έχουμε ε, μαζί με την Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών, μαζί με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να διοργανώσουμε αυτή την κοινή συνάντηση για την κοινή έκθεση που πρόκειται να συντάξουμε εν ώψη της οδηγίας για την ε, ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια των ε, εισηγμένων επιχειρήσεων. Χαίρομαι πολύ που στο πρόγραμμά μας προβλέπεται να μιλήσουν ειδικοί εμπειρογνώμονες για το θέμα και επίσης ε, οι, οι, οι, οι των γνωμοδοτήσεων από τις διάφορες επιτροπές βρίσκονται εδώ και θα λάβουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση από την Επιτροπή των Γυναικών. Στη συνέχεια η κυρία Ρέγνερ θα πάρει το λόγο από την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, από την Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Θα ήθελα να επενθυμίσω εισαγωγικά, γιατί όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, εμεί ήρθαμε να ακούσουμε σήμερα και να λύσουμε τις απορίες μας, να πάρουμε περισσότερα στοιχεία για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα μια ρεαλιστική πρόταση. Οπότε Θέλω απλά να επισημάνω κάποια πράγματα. Από την ε, πλευρά της Επιτροπής των Γυναικών θέλω να επιθυμίσω ότι η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων επιχειρήσεων δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη η Επιτροπή μας έχει συντάξει μια έκθεση σχετική όπου αναδεικνύει όλες τις προκλήσεις της ανέλυξης των γυναικών στην κορυφή των αποφάσεων στις επιχειρήσεις και ε, προτείνει και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μέτρα αποτελεσματικά και δεσμευτικά. Επιπλέον το θέμα αυτό έχει έλθει πολλές φορές σε διάφορα ψηφίσματα ε, και ζητούμε με αφορμή διάφορα θέματα ζητούμε να παρθούν αποτελεσματικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων. Και σας υπενθυμίζω ότι αυτό για μας έχει μια διπλή πηγή έμπνευσης. Από τη μια μεριά είναι η ισότητα των δύο φύλων και η προσπάθεια να την πετύχουμε όπως είναι στις συνθήκες μας και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων καταγεγραμμένο. Από την άλλη πλευρά είναι ένας στόχος για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι έρευνες ευρωπαϊκές και διεθνείς μας λένε τι θετικά αποτελέσματα έχει στις ε, επιδόσεις των επιχειρήσεων, άρα στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Σήμερα λοιπόν η Επιτροπή μας είναι προετοιμασμένη θα έλεγα για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόταση. Θέλουμε όμως να δούμε μαζί με τους ε, εμπειρογνώμονες και μαζί με τα μέλη μας, με τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και με τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων πώς θα ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι για να μπορέσει αυτή η πρόταση να είναι αποτελεσματική. Ήδη στη δική μας έκθεση που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2011 επισημαίνουμε ότι υπάρχουν ανομοιογένειες στο εταιρικό δίκαιο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδα που οι χώρες καταγράφουν ως ποσοστά συμμετοχής στις επιχειρήσεις. Άρα δεν ξεκινάμε από ένα ομοιογενές επίπεδο. Ούτε στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, ούτε και στο σημείο επικίνησης για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών. Και θεωρώ ότι ένα σημείο αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Αν όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε με τους ίδιους τρόπους και το ίδιο χρονικό σημείο, το 2020, το στόχο του 40%. Επίσης θέλω να επισημάνω <clears throat> ποια, ότι είναι σημαντικό για μας ποια είναι η, η εφαρμογή του μέτρου ακριβώς όπως προτείνεται στην οδηγία. Τι είναι πιο σημαντικό και τι υπόκειται στις ε, ε, στις, ε, ε, στις ποινές. Ο στόχος του 40% ή η μη σωστή διαδικασία για να φτάσουμε στο στόχο του 40% συμμετοχής των γυναικών. Επίσης, το άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι προτού φτάσουμε να συζητούμε για μια δεσμευτική πρόταση σήμερα, έχουμε πολύ ασχοληθεί με μεθόδους που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε θελοντικό επίπεδο. Και έχουμε, παρακολουθήσαμε και την προσπάθεια που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προειδοποιήσεις της, με την έγκαιρη ενημέρωση των ε, Προέδρων και Γενικών Διευθυντών για το θέμα αυτό. Είδαμε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά ως προς την ανάληψη των εθελοντικών πρωτοβουλειών. Και επίσης θέλω να επισημάνω Κάτι που ισχυρίζονται κάποια κράτη-μέλη ότι θα μπορούσε να ξεκινήσουμε με μια σύσταση προτού φτάσουμε ή στο νομοθετικό πλαίσιο ότι συστάσεις έχουν ήδη γίνει από το Συμβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη χωρίς αποτέλεσμα. Είμαστε λοιπόν εδώ μπροστά σε μια πρόκληση. Ποια είναι τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε τα αποτελεσματικά και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμοστούν αυτά τα αποτελεσματικά μέτρα. Και η εμπειρία και των δύο επιτροπών και η συμμετοχή και των δύο επιτροπών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων θα συμπλέψουν σε αυτή την πορεία για να έχουμε μια πρόταση που θα έχει αποτελέσματα και θα είναι εφαρμόσιμη στην επικράτεια αυτή όπως είναι σήμερα θα είναι ένα βήμα συμβολικό και ουσιαστικό για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα, για την επίδοση των επιχειρήσεων και για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς η οποία πρέπει να βασίζεται για να είναι αποτελεσματική σε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινού κανόνες και εναρμονισμένα επίπεδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κράτσα για την παρέμβασή σας. Ακούσαμε μία από τις εισηγήτριες. Ακούσαμε την κυρία Κράτσα δηλαδή. Γιατί εδώ έχουμε και εκπροσώπους από την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, όπως ακούσατε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην άλλη εισηγήτρια. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία η πρόταση αυτή την οποία εξετάζουμε είναι ένα δώρο, δώρο προς τις γυναίκες και τους άνδρες για να μπορέσουμε να εντατικοποιήσουμε τη συζήτηση και να επιφέρουμε επικοδομητικά αποτελέσματα για να μπορέσουμε λίγο να ξεπεράσουμε τις παροπίδες οι οποίες υπάρχουν στην ε, κοινωνία με την καλή έννοια βεβαίως και για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε επιτυχημένα το έργο των ε, μεγάλων εισηγμένων εταιριών με την ε, προστίκη, αν θέλετε, περισσότερων ε, διοικητικών στελεχών στα συμβούλια τους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έγινε αυτή η ακρόαση, διότι εδώ θα εξετάσουμε εάν αυτά τα μέτρα, αυτές οι προτάσεις μας επαρκούν, εάν οι κυρώσεις πρέπει να γίνουν ακόμα πιο αυστηρές από αυτές που προβλέπουμε ή, εάν έχουμε το έργο αυτό το οποίο έχουμε αναλάβει ίσως είναι υπερβολικό, ξεπερνάει τα όρια μας. Θα τα εξετάσουμε όλα αυτά λοιπόν σήμερα το απόγευμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει συνεργαστεί πολύ επικοδομητικά, πολύ θετικά με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών, έτσι ώστε να ωφεληθούμε όλοι. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά τις επιχειρήσεις, τους άντρες, τις γυναίκες, τα στελέχη και γενικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιστεύω ότι η συζήτησή μας αυτή θα καταλήξει σε πολύ ενδιαφέροντα ε, και χρήσιμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών, νομικής και επιτροπής δικαιωμάτων των γυναικών. Ε, και θα συνεχίσουμε τώρα, διότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο η εργασία αυτών των δύο επιτροπών, οι στόχοι τους και τα αποτελέσματα συμπεράσματά τους, αλλά και η συμβολή και η συμμετοχή πολλών άλλων ενδιαφερομένων ομάδων και οργανισμών. Ε, ε, αναμένουμε και γνωμοδοτήσεις ε, εδώ στην Επιτροπή μας που συνάδουν με αυτό το, το θέμα. Και τώρα θα ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Όλερ Σμιτ από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αρχίσω ε, <laughs> και να σας δείξω μία φωτογραφία των γκρίζων κοστούμιών των ε, όλων των α, αρένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι όλοι κοστούμαρισμένοι, είναι όλοι κύριοι, είναι όλοι στα γκρίζα. Γιατί σας τα δείχνω αυτό. Διότι θα πρέπει ε, να ξεκινήσουμε τις προσπάθειές μας από τους δικούς μας, από τα δικά μας θεσμικά όργανα, από τα δικά μας ιδρύματα και οργανισμούς. Μπορεί να μου πείτε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση όμως. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό, από μας και ας μην ε, κοροϊδευόμαστε. Πρώτα να, φτιά, να τακτοποιήσουμε το σπίτι μας και μετά τα ενίκο και μετά να δούμε τι μπορεί να γίνει περαιτέρω. Συμφωνώ απολύτως με τους προλαλήσαντες. Συμφωνώ με όλη μου την καρδιά. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο κοινοβούλιο στη δεκαετία, στην πολιτική στη δεκαετία του 70 με την προϋπόθεση ότι όλα λίγο πολύ πρέπει να είναι ίσα, ισότιμα. Πρέπει να υπάρχει ισότητα. Βεβαίω μπορούμε να κάνουμε προτάσεις νομικής φύσεως, αλλά δεν είναι μόνο τα μέτρα, τα νομικά, το, το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, είναι οι νοοτροπίες, οι νοοτροπίες που υπάρχουν. Γι' αυτό θα τονίσω στην έκθεση την οποία θα συντάξω ότι το θέμα είναι πολύ ευρύτερο και δεν καλύπτει δεν αφορά μόνο τα συμβούλια των εισηγμένων εταιρεών. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Αφορά την κοινωνία, το κράτος ε, δικαίου, το ε, κοινωνικό κράτος πρόνοιας. Όταν ήμουνα βουλευτής στη Στοχόλμη πέρασα έξι μήνες μαζί με το γιο μου εθελοντικά. Γιατί το έκανα αυτό, διότι Ήμουν παντρεμένος και ακόμα είμαι και η γυναίκα μου μου είπε «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη από κοινού, ισότητα, έξι μήνες εσύ, έξι μήνες εγώ». Το πιστεύω λοιπόν ακράδαντα. Ε, ε βεβαίως ε, είμαι μετριοπαθή στις απόψεις μου, μετριόφρον. Έχουμε διαφορετικά κοινωνικά συστήματα, διαφορετικά συστήματα προνοίας, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης, ακόμα και στη χώρα μου. Η ερώτησή μου λοιπόν όσον αφορά αυτή την πρόταση είναι ισορροπημένη, είναι αναλογική, είναι ε, σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο το οποίο επιδιώκουμε, είναι εφαρμόσιμη στα κράτη-μέλη. Μήπως αρχίζουμε στο λανσασμένο επίπεδο στις εταιρείε. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε στις χαμηλότερες βαθμίδες των εταιριών αυτών και να ξεκινήσουμε από εκεί την εφαρμογή του μέτρου ισότητας μεταξύ των φύλων. Γι' αυτό στην έκθεσή μου θα τονίσω ιδιαίτερα και ξέρω ότι πολλοί με επικρίνουν, πολλοί δεν συμφωνούν μαζί μου, διότι πολλοί πιστεύουν ότι δεν καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τον, την ομοθεσία πιο αυστηρά. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι αποκρατούσα άποψη. Αν πάει περιπτώσει, αυτή την κριτική την έχω. Εγώ λοιπόν θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να καταλήξουμε σε μία πρόταση η οποία θα συγκρίνεται και με το, με, το Συμβούλιο. Άκουσα ε, φήμες δηλαδή ε, κυκλοφορούν ότι θα μπλοκαριστεί. Υπάρχει μία μειοψηφία η οποία θα μπλοκάρει την πρόταση αυτή. Ε, και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβαστικό κείμενο το οποίο θα είναι αποδεκτό και από τα 27 κράτη-μέλη. Και ε, θα χρειαστεί η πολιτική μας ευελιξία και δεξιότητα για να μπορέσουμε να τα επιτύχουμε πετύχουμε αυτό. Να κάνουμε ένα μικρό συμβιβασμό στα, στις λεπτομέρειες, αλλά ο κεντρικός μας στόχος και η κεντρική μας πορεία να μην αλλάξει. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή δεν θα είναι ευθύνουσα όσον αφορά την προσέγγιση, την προσέγγιση της, θα είναι μία έκθεση η οποία θα αναβαθμίζει την ε, προσέγγιση μας σε όλα αυτά τα θέματα. Και η πρόθεσή μου είναι ταυτόσιμη, είναι ακριβώς ίδια και συμπίπτει 100% με τις απόψεις όλων μας εδώ. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της ΕΚΟΝ και πάμε στην Επιτροπή της Απασχόλησης. Η κυρία Κορνέλσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. I am not a great fan. So wonderful if through self-regulation every... Δεν είμαι υπέρμαχος των ποσοστώσεων και κανένας δεν θα έπρεπε να είναι. Γιατί πιστεύω ότι για να εξασφαλίσουμε την ισότητα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν υποχρεωτικές ε, ποσοστώσει. Αλλά δυστυχώς επί δύο ή τρει δεκαετίες δοκιμάσαμε την αυτορύθμιση και μπορούμε να καταλήξουμε συμπέρασμα ότι δεν δουλεύει. Για λίγους δουλεύει, αλλά για τους περισσότερους όχι. Δεν καταλαβαίνω τις εταιρείε ή τι χώρε που παραπονιούνται ότι πρέπει να δώσουμε τώρα μια ευκαιρία στην αυτορύθμιση. Τη δώσαμε και μάλιστα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά τελικά δεν έπιασε, δεν πόλιασε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι πολλές εταιρείες, πολιτικοί, κυβερνήσεις, πολιτικές ομάδες, όλοι λένε ότι συμφωνούν ότι πρέπει στις διευθυντικές θέσεις να υπάρξουν περισσότερες γυναίκες. Ποτέ δεν είπε κάποιος, όχι, δεν θέλουμε τις γυναίκες εκεί. Όμως, Υπάρχουν τόσες πολλές αντιστάσεις ακόμα. Και όπως ε, είναι διατυπωμένη η πρόταση, αν ένα κράτος έχει μια καλή πολιτική που λειτουργεί και που βοηθάει τις γυναίκες να φτάσουν ψηλά, κανένα πρόβλημα. Αυτό το κράτος δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Αν δεν έχουν όμως μια καλή πολιτική που επιτρέψει τις γυναίκες να φτάσουν εκεί, τότε κάτι πρέπει να κάνουν. Να αρχίσουν να δουλεύουν, να ανασκουμποθούν αλλά το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείε. Αν έχουν μέτρα, ούτω ώστε να επιτύχουν αυτό 40% των γυναικών ε, στις διευθυντικές θέσεις μέχρι το 2020, κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλά, αλλά αν όχι, είναι καιρός να ανασκουμποθούν ήδη από τώρα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν το φόβο που υπάρχει γύρω από αυτή την πρόταση από κάποιους. Η πρόταση φτιάχτηκε για αυτούς που δεν αναλαμβάνουν δράση και όχι για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει πολλά πράγματα ήδη το, το καθήκον μας ως Κοινοβούλιο νομίζω ότι είναι να βελτιώσουμε μαζί την πρόταση. Υπάρχουν κάποιες νομικές αβεβαιότητες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν στη διατύπωση. Πρέπει να συζητήσουμε πώς πρέπει να τη διευρύνουμε, μήπως πρέπει να την κάνουμε πιο σαφή. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα κριτήρια, ε, ποιε χώρε πρέπει να συμμορφωθούν με ποια κριτήρια. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε και μια ευρεία πλειοψηφία γύρω από την πρόταση, όπω είπε και ο κύριος Σμιτ. Πρέπει επίση να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τι λαμβάνει η χώρα στο Συμβούλιο. Και ως πολιτικοί και πολίτες θα πρέπει να βοηθήσουμε ούτω ώστε και στις χώρες μας, στις κυβερνήσεις μας, να σπάσει αυτή η ανασχετική μειοψηφία. Κάτι που πέτυχε ήδη η πρόταση, πριν την ψηφίσουμε ήδη, είναι ότι έθεσε αυτό το θέμα ψηλά στην ατζέντα, προκάλεσε συναισθήματα και νομίζω ότι είναι και καινή ώρα η ισότητα των φίλων να συζητηθεί ξανά. Ευχαριστώ. Και τώρα. Περνάμε στην τελευταία εισηγήτρια γνωμοδοτήσεων, που είναι από την Επιτροπή ΙΜΚΟ, η κυρία Παρβάνουβα. Thank you, President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ως γυναίκα θα μου άρεσε πάρα πολύ να είχα ένα σύζυγο όπως ο Όλε. Ως πολιτικός και μέλος της Επιτροπής θα ήθελα να έχουμε ένα συμβούλιο το οποίο να λέει θα υπάρξουν ίσες ευκαιρίες άνδρων και γυναικών και δεν συζητείται αυτό. Αλλά έτσι όπως έχει η κατάσταση, όλες οι, όλοι οι συνάδελφοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους. Ούτε σε 20, ούτε σε 30 χρόνια, ούτε σε 20 αιώνες, ούτε σε 30 αιώνες δεν πρόκειται να φτάσει η αυτορύθμιση για να πετύχουμε το αποτέλεσμα το που θέλουμε. Σίγουρα λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε και άλλες εναλλακτικέ πέραν των επιλογών που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω το εξή: Όποια και αν είναι η σύνθεση των θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνώ απολύτω με τον Όλε Σμιτ. Πρέπει ε, να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μα αργά ή γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προβληματιστούμε για ε, το κλάδο των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα 3 τέταρτα των πολιτών είναι υπέρ των ποσοστώσεων και 49%, δηλαδή σχεδόν το μισό, είναι υπέρ των χρηματικών προστήμων ως ε, ο πιο κατάλληλος μηχανισμός για τη θέση σε ισχύ και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Αυτό δείχνουν οι έρευνες. Είναι λογικές αυτές οι προσδοκίε. Οι πολίτες πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ισότητα των φύλων και δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ούτε άλλος τρόπος. Ω εισηγήτρια λοιπόν τη γνωμοδότηση για την εσωτερική αγορά, προσπάθησα να καταλήξω σε ένα ισορροπημένο κείμενο για τη λειτουργία της ε, εσωτερικής αγοράς, για τη νομική βεβαιότητα, για τις επιχειρήσεις, νομική ασφάλεια και ε, για το ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των καταναλωτών κατά τη λήψη αποφάσεων στα διοικητικά συμβούλια. Το 70% των αποφάσεων που έχουν να κάνουν με την καταναλωτική δαπάνη λαμβάνεται από γυναίκες. Άρα αν είναι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια θα δώσουν πληροφορίε εκ των έσω για τις, για τις επιλογές του καταναλωτή και νομική ασφάλεια θα υπάρξει και στις ε, επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περισσότερα του ενός κράτη-μέλη. Ε, δυστυχώς μέχρι σήμερα υπάρχει κακοφωνία ως προς τα διοικητικά συμβούλια σε όλη την Ένωση. Αυτή η διαφοροποίηση έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Οι επιχειρήσεις με διασυνοριακή λειτουργία και δραστηριότητα χρειάζονται ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο, σταθερό, βέβαιο, για να υποφεληθούν από την πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Ε, το φαντάζεστε άλλωστε, αν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες, δεν ξέρει τελικά ε, ποια ε, νομοθεσία θα ισχύσει για τις δραστηριότητες της ε, στην άλλη χώρα και το καθεξής. Σύμφωνα με τη μελέτη της McKinsey, McKinsey οι οικονομικές επιδόσεις και η κερδοφορία των επιχειρήσεων αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ίση εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια. Επομένως, η ε, όλα αυτά συνδέονται όχι μόνο με την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης, αλλά θα έχει θετικό αντίκτυπο και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Και θα ήθελα να πω ότι σε καιρούς οικονομικής κοινωνικής, χρηματοπιστητικής αλλά και δημογραφικής κρίσης είναι σπατάλη ανθρωπίνων κεφαλαίων να μην χρησιμοποιείτε και να μην αξιοποιείτε το ίμιση του πληθυσμού. Παρόλο που υπάρχουν στοιχεία ότι η συνεισφορά ε, των γυναικών είναι εξαιρετικά πολύτιμη και θετική. Τίποτα δεν δείχνει ότι οι περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια βλάπτει. Αντιθέτως, ε, οδηγεί σε Μία 10% αύξηση της εκπροσώπησης γυναικών στα διοικητικά συμβούλια οδηγεί σε 20% αύξηση των εισοδημάτων, των εσόδων μιας επιχείρησης και καμία μελέτη δεν δείχνει ε, αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι σαφέστατο. Και σύνθεση άλλη, ε, στο κείμενό μου προσπάθησα να συμπεριλάβω πρωτοβουλίες και κίνητρα για τα κράτη-μέλη, ε, να ενθαρρύνω ώστε να έχουμε αναφορές για το τι πρόοδος έχει επιτευχθεί, ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στο τομέα αυτό και για να διευκολυνθεί και η πρόσβαση των γυναικών σε επιχειρηματικά δίκτυα. Θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν την πολιτική τους για τους ανθρώπινους πόρους για να στηρίξουν το ταλέντο των γυναικών. Και αυτή θα είναι η θέση ε, που θα εκφραστεί στη γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε ακούσει τις ε, δύο εισηγήτριες. Μετά ακούσαμε ε, τους εισηγητές που θα έχουν ε, γνωμοδοτήσεις. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Σάρμα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Θα μας πει για το περιεχόμενο της παρέμβασής της. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Να σας πω ότι δεν μιλούμε για ποσοστώσεις και το σημαντικό είναι να μην περδέψουμε τα πράγματα. Η ποσόστοση έχει αρνητική χρειά και προκαλεί έντονα συναισθήματα. Δεν μιλούμε λοιπόν για ποσοστώσεις, μιλούμε για ε, ε στοχευμένους σκοπούς, ο targeted objectives, ότι δηλαδή αυτός είναι ένας στόχος τον οποίο θέλουμε να επιδιώξουμε. Δεν υπάρχει πολιτή στον κόσμο που να μην έχει στόχο. Οι εταιρείε δίνουν στους πολιτές τους στόχους γιατί πρέπει οι στόχοι να επιτυχάνονται και είναι σημαντικό να έχουμε αυτού τους ε, στόχους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ τα εμπρός. Η νοοτροπία και η πραγματικότητα είναι η εξή. Είχαμε αυτορύθμιση για αιώνε και δεν έχει ε, σημειωθεί καμία αλλαγή η πίεση και το γεγονός και μόνο το ότι συζητούμε αυτή την οδηγία έχουν προκαλέσει κινήσεις σε διάφορες χώρες, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στη Δανία. Σημειώνονται ριζοσπαστικές αλλαγές και μόνο επειδή συζητείται το θέμα, χωρίς τίποτα άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να το σπρώξουμε ακόμα περισσότερο, να το πιέσουμε. 24 ε, επιχειρήσεις υπέγραψαν τη δέσμευση και μεγάλο ποσοστό ε, εξ αυτών ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν δεν προβάλλεται επιχειρήματα, τότε αυτά δεν τα ακούει ο επιχειρηματικός κλάδος του οποίου εγώ είμαι μέλος. Κανένα συγκεκριμένο επιχείρημα δεν έχει προβληθεί πουθενά το οποίο να λέει ότι αυτό δεν είναι καλό για τις business και τις επιχειρήσεις γενικότερα. Οι μη εκτελεστικοί διευθύνοντες υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητοι από την εταιρεία. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να ξέρουν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των προτέρων και να μην έχουν γνώση τη εταιρεία εκ των προτέρων. Και οι περισσότεροι διορίζουν κάποιον που ξέρουν, κάποιον που γνωρίζουν όταν πρόκειται για άντρα. Όμως οι γυναίκες που διορίζονται ως μη εκτελεστικές διευθύνουσες σύμβουλοι είναι πραγματικά ανεξάρτητες και θεωρούνται οι άνδρες ως εξαιρετικών προσόντων. Όμως ε, τις γυναίκες τις βάζουμε στο στερεότυπο ότι είναι οι χρυσές φούστες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτό το στερεότυπο. Τύπο. Πράγματι, πολλές γυναίκες έχουν περισσότερες από μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό όμως συμβαίνει και με τους άνδρες. Και το γεγονός είναι ότι παραμένουν οι πολύ περισσότεροι άνδρε που έχουν διάφορε θέσει ω μέλη σε διοικητικά συμβούλια χωρί να έχουν δουλειά, να, καμία άλλη δουλειά να μην κάνουν. Ενώ οι γυναίκε μπορεί να τι έχουν, αλλά έχουν και θέση απασχόληση. Δουλεύουν σύν τη άλλη. Έχουν ίσα προσόντα ή ίσες ε, δυνατότητε, δεξιότητε και μάλιστα είναι και νεότερε. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε νορβηγική μελέτη. Άρα Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε και ε, τα ευρήματα της ε, μελέτης συνηγορούν προς το αυτό. Είναι οικονομικό το θέμα να έχουμε περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Δεν είναι θέμα φύλου. Εκεί όπου υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια έχουμε περισσότερη διαφάνεια, έχουμε αύξηση στην τιμή της, εποχής και, της μετοχής και έχουμε αύξηση ε, της απόδοσης της επένδυσης, του λόγου αυτού δηλαδή, του ρόη δεν υπάρχει επιχείρημα κατά και θέλω να το στηρίξω αυτό, να το ε, πιέσουμε να γίνει όσο να το περισσότερο. Στηρίζω τις δύο εισηγήτριες, να στηρίξουμε όλοι μαζί την κυρία Ρέντιν για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα θα συνεχίσουμε και θα Με το θεσμικό φορέα ο οποίος, για το πούμε έτσι, ξεκίνησε όλα αυτά τα θέματα. Η κυρία Τσιομπάνου Ντοντέα από την Κομισιόν. Ο, κύριος να έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση με τους συναδέλφους σας. Εάν κατάλαβα καλά, ε, άκουσα από την, ε, τους διερμηνείς ε, βεβαίως ότι ε, στην καρδιά όλης αυτής της συζήτησης είναι το θεσμικό όργανο στο οποίο είμαι εγώ. Η Κομισιόν είναι η οποία ξεκίνησε και βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών των προτάσεων. Η πρόταση αυτή γιατί ε, έχει ένα, μια ιστορία. Θα σας αναφέρω λοιπόν πώς προέκυψε πριν, πριν αναφερθώ σε ορισμένα, σε συγκεκριμένα στοιχεία. Ε, αναπτύχθηκε η πρόταση αυτή μέσα σε ένα πλαίσιο ε, μετα, συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και πολλών εταιριών που εδραίωσαν πολιτικές και συγκεκριμένες και υλοποίησαν συγκεκριμένα μέτρα για να ενθαρρύνουν και αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα. Αυτή η προσπάθεια εφαρμόστηκε και στην εκπαίδευση ε, ε, και γενικά ωφέλησε και πολλούς άλλους τομείς της ε, κοινωνικής ζωής. Παρόλο που υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, Έχουμε δει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένους δείκτες ε, μετρήσιμους με τους οποίους μπορούμε να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από τις αγορές από τον Οκτώβριο πέρσι δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή μόνο 15,8% γυναικών είναι μέλη, ε, έχουν εκτελεστικές θέσεις στα διοικητικά συμβούλια εταιρεών και 16 μόνο, 16,8% στα διοικητικά συμβούλια είναι γυναίκες. Από τότε που έχουμε τα στοιχεία αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, η πρόοδος που σημειώθηκε ήταν ελάχιστη 0,8-0,9% ετησίως. Ε, αυξήθηκαν αυτά τα ποσοστά. Αυτά δείχνουν ότι η αντίδραση σε, αυτέ αυτές τις προτάσεις ήταν ανεπαρκής και το Συμβούλιο το 93-94 πρότεινε θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών. Το 93 το Συμβούλιο αναθεώρησε το θέμα αυτό και εξέδωσε μία σύσταση στα κρατημέλη για να λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν τη συμμετοχή των γυναικών στις οικονομικές λήψεις αποφάσεων. Δηλαδή πολύ πιο συγκεκριμένη σύσταση. Και πριν από δύο χρόνια, την άνοιξη του 2011, η Αντιπρόεδρος κυρία Ρέντιν υπέβαλε την δική της πρόταση προς τον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία ε, πρόταση η οποία είχε μία θα έλεγα αντίδραση που πολύ χαμηλών τόνων από τις επιχειρήσεις. Στο μεσοδιάστημα είδαμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ένας περιορισμένος αριθμό κρατών μελών ανέλαβαν ορισμένες πρωτοβουλίες, ε, είτε μέσα στην νομοθεσία, με νομοθετικά μέτρα, είτε με αυτορύθμιση και άλλες πρωτοβουλίες. Αλλά η απόδοση, το αποτέλεσμα σε όλη την Ένωση είναι πολύ ανομοιογενές. Από 4% συμμετοχή δηλαδή γυναικών σε 26 20, μέχρι 29% ή λίγο παραπάνω από 30% συμμετοχή γενικών στα διοικητικά συμβούλια που είναι εταιρεών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Ε, πολύ ανομοιογενή λοιπόν τα αποτελέσματα. Γι' αυτό ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει και από αυτή την οπτική γωνιά πρέπει να εξετάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής, Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής Επιτροπής και γι' αυτό η Κομισιόν έχει υποβάλει μια πρόταση η οποία είναι φιλόδοξη, ρεαλιστική και ανάλογη, έχει μια ε, αναλογικότητα με αυτά τα οποία επιζητούμε. Είναι φιλόδοξη διότι στοχεύει σε έναν γενικό στόχο 40% μέχρι το τέλος της δεκαετίας συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου ε, στις, ε, στα διοικητικά συμβούλια συγμένων εταιριών. Αυτό σημαίνει ότι ε, είναι η, διάσταση του φίλου αντιμετωπίζεται ισότιμα. Εάν υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες, τότε πρέπει να αυξηθούν 40%. Αν υποεκπροσωπούνται οι άνδρες σε πολύ ελάχιστους κλάδους βεβαίως, αλλά υπάρχει, υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα όπου υποεκπροσωπούνται λοιπόν οι άνδρες και εκεί πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό. Κυρίως όμως οι προτάσεις αυτές ε, και οι δικαιούχοι, οι ωφελούμενοι από αυτές από την πρόταση είναι οι γυναίκες. Βεβαίως η κατάσταση αυτή εξαρτάται και από το καθεστώς ιδιοκτησίας των εταιριών αυτών. 20, ε, το 2020 είναι η προθεσμία για τις ε, εταιρείες γενικώ, αλλά ε, γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και στις δημόσιες επιχειρήσεις ο στόχος είναι πιο ε, φιλόδοξος και το, η προθεσμία έχει οριστεί το 2018. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε πιο φιλόδοξοι και δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε, σε ένα τυφλό ε, ποσοστό, σε ένα τυφλό νούμερο ποσοστώσεων, διότι αυτό δεν είναι ικανοποιητικό και δεν θα λύσει τα προβλήματα σε, ένα διοικητικό συμβούλιο του υποεκπροσωπούμενου φίλου. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι τα προσόντα, οι δεξιότητες και το ταλέντο ενός υποψηφίου ή μίας υποψηφίου είναι το καθαριστικό στοιχείο. Βάσει αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Υποπτικά Συμβούλια θα αποφασίσουν αν είναι κατάλληλος ο, ή υποψήφια ε, για τη θέση. Αλλά θα πρέπει ακριβώς σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συνεχεία υπό ίσες συνθήκες να δίνεται προτεραιότητα στον υποψήφιο εκείνον ο οποίος ανήκει στο υποεκπροσωπούμενο φύλλο. Προϋπόθεση όμως για την τελική επιλογή αποτελούν οι, οι, οι, ίδιες συνθήκες όσον αφορά ε, τα προσόντα και τις δεξιότητες. Δεν είναι λοιπόν μόνο τα οι ποσοτικοί στόχοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ε, ε μας ενδιαφέρουν μέχρι το 2018. Θέλουμε πέραν των ποσοτικών στόχων να εδραιώσουμε μία διαρκή ε, διαδικασία, μία ε, προσέγγιση για το μέλλον που θα παράγει αποτελέσματα και μετά τον, τη χρονολογία αυτή μετά από το 2028 όταν θα εκπνεύσει αυτή η οδηγία. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να παγιώσουμε, να εδραιώσουμε μια αντίληψη, μια προσέγγιση και πέραν αυτών των ημερομηνιών. Και η πρόταση αυτή τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να καθιερωθούν διαφανείς συνθήκες προσλήψεων διαφανείς αντικειμενικές και με τρεις συγκρίσιμες συνθήκες προσλήψεων, συγκρίσιμα κριτήρια μάλλον προσλήψεων. Έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και τις διαφορετικές, ε, τις ιδιαιτερότητες που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Άλλα κράτη, μερικά κράτη τα οποία είναι πιο φιλόδοξα έχουν θέσει ενισχύ ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Πρέπει να αποδείξουν όμως ότι πράγματι έχουν επιτευχθεί αυτά τα αποτελέσματα και στην Κομισιόν αλλά και δημόσια. Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις επιτρέπουν στα φιλόδοξα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν το σύστημά τους και να είναι εφαρμόσιμο, να λειτουργεί. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο αναστέλλεται η οδηγία για αυτά τα κράτη-μέλη και θα εφαρμοστεί, θα τεθεί πλήρως ενισχύ μόνο εάν τα αποτελέσματα δεν είναι, αυτά τα, δεν είναι τα επιδιωκόμενα. Και το τρίτο χαρακτηριστικό που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτή την πρόταση νομοθετικής φύσεως είναι η αναλογικότητα. Και το χαρακτηριστικό ότι είναι η κατάλληλη πρόταση για τις κατάλληλες συνθήκες και για τους κατάλληλους στόχους. Αυτό το, το βασικό επιχείρημα που στηρίζει αυτό το στόχο είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά διοικητικά συμβούλια και διαφορετικά μέλη στα διοικητικά συμβούλια. Υπάρχουν μέλη τα οποία έχουν εποπτικό καθήκοντα, εκτελεστικά καθήκοντα και μη εκτελεστικά καθήκοντα. Η στόχη για το 2020, αυτό το 40% αναφέρεται συγκεκριμένα στα μέλη των συμβουλίων, των εποπτικών συμβουλίων. Όμως, Ζητούμε τα, κράτη-μέλη να υποχρεώσουν τις εταιρείες να μας παρουσιάσουν τους δικούς τους στόχους όσον αφορά την ισόρροπη συμμετοχή των φίλων στα διοικητικά συμβούλια η πρόταση αυτή σίγουρα δεν καλύπτει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι επειδή θα επιφέρει μεγαλύτερο βάρος στις μικρομεσαίες, αλλά επειδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν χαρακτηριστικά τα οποία δεν συνάδουν με την πρόταση αυτή. Είναι μικρές επιχειρήσεις, συνήθως κονιακές, και έχουν ένα περιορισμένο δυναμικό όσον αφορά την οργάνωση μιας ε, διαφανούς και αντικειμενικής ε, διαδικασίας προσλήψεων. Επίσης η πρόταση αυτή δεν καλύπτει δεν καλύπτει ορισμένου οικονομικού τομεί, εκτό αν το κράτο μάλιστα επισημεί αντίθετα. Λοιπόν, δεν καλύπτει Α, τα, το, το υποεκπροσωπούμενο φύλλο σε περιπτώσεις όπου αυτή η ε, μικρή εκπροσώπηση είναι κάτω του 10% σε μια επιχείρηση. Επίσης προσπαθήσαμε να, οι προτάσεις μας να είναι αναλογικές στις διατάξεις περί κυρώσεων. Ορισμένοι μας έχουν επικρίνει επειδή δεν έχουμε προτείνει αυστηρές ή και ποινικέ κυρώσεις. Εμείς προσπαθήσαμε να, ε, να, να, συνάδουν οι, προτάσεις μας με τα πρότυπα, ε, ε, με τα, τα πρότυπα των προστήμων και των ποινών που ορίζονται σε άλλες οδηγίες. Ε, τώρα θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι κυρώσεις ε, που επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη να είναι αναλογικές ε, όσον αφορά και τους άλλους τομείς. Γιατί, διότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια, είναι δική τους ευθύνη να ε, ορίσουν ε, ποινές, πρόστιμα και κυρώσεις ανάλογα με τη μορφή και το μέγεθος της εταιρείας θα πρέπει λοιπόν η παραβίαση αυτών των κανόνων να, να εμπίπτει μέσα στο γενικό πλαίσιο ε, παραβιάσεων και επιβολής κυρώσεων του, του κράτους μέλους. Επίσης επιδιώκουμε την αναλογικότητα όσον αφορά την εποπτεία και ε, την ε, σύνταξη εκθέσεων αναφοράς ε, των εταιριών αυτών μέχρι το 2028. Οπότε έχουμε ακριβώς αυτή τη ρήτρα κατάληξης της οδηγίας. Ε, θέλουμε κύριε Πρόεδρε όλη αυτή η νομοθετική πρόταση να είναι ε, αναλογική, να είναι ισορροπημένη, ε, να βασίζεται σε δυνατά επιχειρήματα και να καταλήξει στο επιδιακόμενο αποτέλεσμα που είναι η επιβολή και η παγίωση της ισότητας των φύλων. Πιστεύω ότι όλες αυτές μας οι προσπάθειες είναι παράλληλες και συμφωνούν απόλυτα με τους δικούς σας στόχους. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Και τώρα... Τελειώσαμε την εισαγωγική φάση και περνάμε στο πρώτο πάνελ, στο πρώτο τμήμα του εργαστηρίου μας. Ακούσαμε τώρα ποια είναι τα βασικά θέματα. Και θα πάμε λοιπόν στο πρώτο πάνελ που απαρτίζεται από δύο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό της παρουσίας των γυναικών σε ανώτατα, ανώτατες θέσεις, ανώτατες δικές θέσεις. Είναι η Κολέτ Φάγκαν και η Σίλβια Γκόμες Ανσόν. Χαίρομαι πολύ που είσαστε παρούσα. Ευχαριστώ που με καλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Να το όνομά μου. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο ε, είναι η βάση ε, πάνω στην οποία στηριχθήκαμε. Στηριχθήκε η έρευνά μας. Ε, η έρευνά μας εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια με δύο τρόπους ξεκινήσαμε με μία ε, διεθνή ε, επισκόπηση. Θα μιλήσει για αυτή η συναδελφός μου Σίλβια Γκόμες Ανσόν και ε, περιλαμβάνουμε 8 περιπτωσιολογικές μελέτες από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε τρεις σκανδιναβικές χώρες με μεγάλη ιστορία συγκεκριμένων θέσεων στα διοικητικά συμβούλια. Έχουν ούτως ή άλλως χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ποσοστώσεις στο Δημόσιο βίο. στα διοικητικά συμβούλια. Ε, εν συνεχεία μίλησαν για ποσοστώσεις σε ιδιωτικές εταιρείες. Η Ισπανία και η Γαλλία πιο πρόσφατα υιοθέτησαν ε, τις ποσοστώσεις. Η Ισπανία το 2007 με 8 ετή ορίζοντα, 40% ε, ήταν ο στόχος. Η Γαλλία ε, είχε δώσει έναν εξαετή ορίζοντα για να φτάσει το 40%. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήθελε παρέμβαση, παρότι επέβαλε στόχους επιτυχώς ως κίνητρο ας πούμε για να τοποθετηθούν γυναίκες σε ανώτατες θέσεις. Και το 2011 με την έκθεση Davis ε, μπήκαν οι στόχοι, ε, συνεχεία έγιναν κάποιες έρευνες από τις ε, εταιρείε και ορισμένες εταιρείε ε, υπέραψαν μια δέσμευση ότι θα σεβαστούν το στόχο και δεν θα έχουν μόνο άντρες σε θέσεις διοικητικές. Η Σλοβενία και η Ουγγαρία έχουν μια μακρά παράδοση ισότητας ε, των φύλων που την ε, κληρονόμησαν και την προώθησαν μετά με την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν χρησιμοποιούν στόχους ή ποσοστώσεις ε, για να υπάρξουν θέσεις, ανώτατες διοικητικές θέσεις. Γενικά, έχουμε τρία είδη εθνικών πολιτικών με τα οποία λειτουργούν οι χώρες. Καταρχάς, η μη παρέμβαση. Η ιδέα ότι το αφήνει στα άτομα να αποκτήσουν γνώσεις, ζήλο, να προχωρήσουν και στις οργανώσεις, ούτω ώστε να έχουν εσωτερικούς δείχτες για τις επιδόσεις και αργότερα υποτίθεται ότι η χώρα θα παίξει το ρόλο της, γιατί αυτά τα πράγματα λειτουργούν αλυσιδωτά. Διάφοροι ε, ερευνητέ η Μάντι Σάρμα ε, ερεύνησαν αυτά τα πράγματα, αλλά γενικά στην Ευρώπη έχουμε περίπου ε, το 1 τρίτο των θέσεων που το έχουν οι γυναίκες, έχουμε το 50% των επαγγελματικών θέσεων που έχουν οι γυναίκες, επομένως υπάρχει, υπάρχουν στοιχεία Τώρα, υπάρχουν συστάσεις ήπιας νομοθεσίας σε διάφορες χώρες. Εδώ τίθενται στόχοι, εξηγούμε ας πούμε τους στόχους και συνεχεία έχουμε νομοθεσία. Αξιοκρατικές ε, ποσοστώσεις. Ε, μερικές φορές ε, εδώ δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ακριβώς ε, ή αξιοκρατικός διορισμός. Τι προέκυψε από την ερευνά μας. Ορισμένα δεν μας εντυπωσιάσουν. Οι ποσοστώσεις, καλοσχεδιασμένες ποσοστώσεις ή η απειλή των ποσοστώσεων, όπως έκανε η Σουηδία, η οποία απειλή θα κάνει αυτό που έκανε η Νορβηγία, ε, βοήθησε στο να βελτιωθεί η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις. Ε, και αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική ζωή. Οι κυβερνητικές οι κυβερνητικοί κώδικες ε, είναι λιγότερο αποτελεσματικοί, είναι, έχουν συμβολική σημασία, αλλά στις αιτήσιες εκθέσεις απλώς τους ρίχνουμε μια ματιά και τους αγνοούμε τους κώδικες αυτούς. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες βέβαια και αυτό τι σημαίνει. Ότι όλα εξαρτώνται από την ποιότητα του εργαλείου και από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εισάγεται. Από την εκάστοτε συγκυρία δηλαδή. Θα πρέπει να έχουμε ας πούμε σωστές προθεσμίες εφαρμογής, θα πρέπει να δούμε το επίπεδο και το είδος των κυρώσεων, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει εμπειρία, κατανόηση των στόχων, των ποσοστώσεων ή των σχεδίων δράσης για την εισόδο των φύλων αν υπάρχουν διαφορές τομεακές, αν υπάρχουν τομείς όπου κυριαρχούν ας πούμε, οι άντρες, όπως ας πούμε, τα ορυχεία και η εξόριξη, και όπου είναι δύσκολο ας πούμε, να βρει γυναίκες, ή επιστημονική κλάδη, ή ο οικονομικός και χρηματοπιστωτικός κλάδος, όπου τώρα πια το 50% είναι γυναίκες. Αυτό είναι στο διαφορά το σχεδιασμό. Τώρα, ε, συντρέχουν λόγοι. Ποια είναι τα επιχειρήματα. Η Σίλβια θα μιλήσει πιο λεπτομερώς γι' αυτό. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι με βάση την βιβλιογραφία υπάρχουν λόγοι για να υπάρχει διαφοροποίηση ε, και ισορροπία ανδρών και γυναικών. Γιατί είναι η, η παραγωγικότητα είναι καλύτερη, ε, υπάρχει διαφορετική επικοινωνιακή επίδοση ανδρών και γυναικών, άλλη προσέγγιση των δύο φύλων κτλ. Επίσης ε, σπάνε τα στεγανά ε, που οφείλονται στα φύλλα κτλ. Τώρα, αν πούμε, ας δούμε τα διοικητικά συμβούλια. Αν δούμε, ας πούμε, 12 άτομα που απαρτίζονται, 12 άτομα απαρτίζουν, ας πούμε, το, Διοικητικό Συμβούλιο, πώς θα πάνε, ποιε είναι οι επιδόσεις τους, ε, η αποτελεσματικότητά του. Τότε είναι δύσκολο να, δούμε, να, να βρούμε στοιχεία. Υπάρχουν πολύ λίγε αποδείξει ε, αποδείξεις, για να που δείχνει ότι οι επιδόσεις είναι χειρότερες ε, από την ισότητα των φίλων. Υπάρχουν λίγες μελέτες, αλλά όλο και περισσότερες αυξάνονται, ας πούμε. Χρειαζόμαστε μια για πιο μεγάλη χρονική περίοδο για να συλλέξουμε αυτές τις ε, αποδείξεις. Να σας πω κάποια στοιχεία παρόλα αυτά. Μερικοί λένε που είναι κατά των ποσοστώσεων και αναφέρουν την περίπτωση της Νορβηγίας. Ε, λένε ότι οι βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, ας πούμε, είναι χειρότερες ε, όταν επιβάλλουμε τις ποσοστώσεις. Υπάρχουν δύο λόγοι ίσως. Όταν, ας πούμε, έχετε ανακατατάξεις έτσι, σε μια ομάδα. Ε, η ομάδα πρέπει να γνωριστεί για να αποδώσει. Αν ας πούμε χάσεις πέντε άντρε από ένα συμβούλιο και φέρεις πέντε νέους, θα πρέπει πρώτα να καταλαγιάσει το πράγμα, να ομαδοποιηθεί, να υπάρξει μια ομάδα μάλλον, μια δυναμική ομάδας. Επίσης, υπάρχουν προκαταλήψεις ε, από επενδυτές μερικές φορές. Α, τι κάνετε αυτή. Η εταιρεία έφερε γυναίκες ας πούμε. Ε, έφερε γυναίκες και ε, θεωρούν ότι οι επιδόσεις της εταιρείας αυτής θα είναι χειρότερες. Ε, χάνουν την εμπιστοσύνη αλλά αυτό γίνεται βραχυπρόθεσμα. Επίσης το 2012 έγινε μια μελέτη ε, στην Ελβετία για εταιρείε στην Ελβετία που είδε ότι οι ίδιες εταιρείες του ίδιου κλάδου ε, για μία περίοδο έξι χρόνων, όταν είχαν τουλάχιστον μία γυναίκα σε διοικητικά συμβούλια, πήγαν πολύ καλύτερα σε επιδο... είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις. Και ακόμα και μέσα στην περίοδο της ε, οικονομικής κρίσης. Επομένως, το επιχείρημά μου είναι... Με βάση τα στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καταστροφικό, είναι καλό για τις επιχειρήσεις να έχουμε γυναίκες ε, στα δουσού και με αυτόν τον τρόπο προσλαμβάνουμε ε, από ευρύτερη ε, βάση παρά να παίρνουμε μόνο συμβολικά ας πούμε γυναίκες. Καλό είναι να έχουμε ένα ε, ευρύτερο πουλ από το οποίο προσλαμβάνουμε. Φυσικά οι ποσοστώσεις είναι επίμαχες. Το βασικό είναι τι αντιλήψεις έχουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τα θέματα της δικαιοσύνης, της ικανότητας, της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Μερικές φορές δεν ξέρουμε αν μπορούμε να προσλάβουμε, αν έχει νόημα να κάνουμε διακρίσεις. Μερικές φορές ε, λέμε τι πρέπει να προωθήσουμε, την αυτονομία των επιχειρήσεων ή τη λογοδοσία απέναντι στην κοινωνία. Τώρα, αν χρησιμοποιεί ε, ούτως ή άλλως στη χώρα σου ή γενικά στις επιχειρήσεις της χώρας σου τις ποσοστώσεις, είναι κάτι που το έχουμε αφομοιώσει, το έχουμε μάθει. Ε, Παραδείγματος χάρη, στην, όταν υπάρχει μια παράδοση, σε μια χώρα ε, είναι κάτι που το έχει αφομοιώσει και επομένω, ούτω ή άλλω μπορεί να χρησιμοποιήσεις αυτή την ε, εμπειρία καλύτερα. Μαθαίνουμε καθώς προσπαθούμε. Το βασικό είναι επίσης ε, πώς προωθούνται αυτές οι πολιτικές, τι επικοινωνία υπάρχει γύρω από αυτές. Επίσης, ποιο είναι το πλαίσιο με στο οποίο το επιβάλλουμε. Παραδείγματο χάρη, η καναδική εμπειρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, δημιουργήθηκε μια δέσμη κριτηρίων ικανότητας. Δηλαδή, κοιτάς παραδείγματο χάρη τι ικανότητε έχουν οι άνθρωποι που έχει ένα διοικητικό συμβούλιο και τι σου λείπει, ούτως ώστε να το ψάξεις. Τα συμπεράσματά μου. Η αποτελεσματικότητα των ποσοστώσεων και των στόχων απαιτεί ε, μια ευρύτερη δέσμη μέτρων ισότητας. Οι κανονισμοί έχουν, ε, δεν έχουν πολλές, ε, πολλή επιτυχία. Οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις γενικά είναι πιο αποτελεσματικές από τα θελοντικά μέτρα, παρότι ένα plan B θα μπορούσε να είναι στόχος, δέσμευση και έλεγχος. Ε, εδώ στον Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το Plan B μας ε, οδήγησε σε κάποιες αλλαγές. Θα μιλήσουν για αυτό το θέμα και άλλοι ομιλητές. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική επικοινωνία, να μιλήσουμε αποτελεσματικά για τα νέα μέτρα. Πρέπει να αμφισβητήσουμε επίσης ε, την καθεστική αντίληψη και πρέπει να υπάρχουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για κάθε παρέμβαση. Πρέπει να δώσουμε μια συγκεκριμένη προθεσμία, μάλλον λογική προθεσμία, πάτηματος χάρη. Ε, σε ένα διοικητικό συμβούλιο στο Ενωμένο Βασίλειο έχεις 12 εκτελεστικές διευθυντικές θέσεις και 6 μη εκτελεστικές. Ε, επομένως, για να κάνουμε οποιοδήποτε αλλαγές χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να πετύχουν. Επίσης, οι έρευνες που κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες ε, παίζουν σημαντικό ρόλο. Χρειάζεται κάποιος χρόνος για να δημιουργηθεί ε, μια ομάδα ανθρώπων από την οποία μπορούν να αντλήσουν όταν υπάρξουν και θέσεις. Εγώ είμαι σε ένα διοικητικό συμβούλιο και όπως και η κυρία Σάρμα ε, χρησιμοποιούμε δείχτες, μας βοηθούν αυτοί, ούτως ώστε να εστιάσουμε. Επίσης έχουμε και στόχους για την διαφοροποιημένη συμμετοχή άντρων και γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που δεν σας παρουσίασα, κοιτούσα προς τα δεξιά και εσείς βρισκόσασταν στα αριστερά. Ε, θα έπρεπε λόγω παρελθόντων μου να το είχα καταλάβει, γι' αυτό δεν έκανα σωστή ε, ε, σύσταση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν καθηγήτρια κυρία Φάγκαν Είστε καθηγήτρια κοινωνιολογίας και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεισφορά σας. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην καθηγήτρια κυρία Σίλβια Γκόμας Ανσόν, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Οβιέδο της Ισπανίας για θέματα ε, χρηματοοικονομικά και λογιστικής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Είναι χαρά για μένα που μπορώ να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Αν δεν σας πειράζει, θα ήθελα να μιλήσω στα ισπανικά, παρόλο που οι διαφάνειες είναι στα αγγλικά. Στόχος της παρουσίασής μου είναι, κατά κύριο λόγο, να αναφερθώ στις οικονομικές επιπτώσεις που έχει η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εισηγμένες. Όπως ήδη έχουμε παρουσιάσει εδώ, ε, παρατηρούμε την εξέλιξη της παρουσίας των γυναικών στις εισηγμένες επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Και η εξέλιξη αυτή ήταν εξαιρετικά μειωμένη. Η παρουσία δηλαδή των γυναικών ήταν μειωμένη και η αύξησή τους ήταν, δεν ξεπερνούσε το 0,5 ή 0,8% ετησίως. Αν αναλύσουμε όμως την ε, παρουσία γυναικών ως προέδρων ε, των μεγάλων εισηγμένων επιχειρήσεων, τότε το ποσοστό είναι ακόμα μικρότερο, 3% και όχι 10% και αυξήθηκε μόνο 1% μέσα σε 10 χρόνια. Τούτων λεχθέντων, η Ευρώπη είναι η ήπειρο όπου η παρουσία των γυναικών στα ΔΣ είναι αυξημένη σε σχέση με τι υπόλοιπε χώρε. και αυτό οφείλεται στη θέσπιση ποσοστώσεων σε ορισμένε χώρε για την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Πολλέ είναι οι διαφορές μεταξύ χωρών. Έχουμε τι σκανδιναβικέ χώρε και έχουμε τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, εκεί παρατηρούμε και στις δύο αυτές περιοχές μεγαλύτερη παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, ενώ στις μεσογειακές χώρες η παρουσία των γυναικών είναι κατά πολύ μειωμένη συγκριτικά. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι το ίδιο να εξετάζουμε μια γραφική παράσταση που παρουσιάζει τα ποσοστά των γυναικών στα ΔΣ, όσα να ήταν μια ε, συγκεκριμένη ε, γραφική παράσταση με πολύ συγκεκριμένες ε, επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχουν και άλλες τόσες και πολύ περισσότερες όπου δεν μπορεί να μην υπάρχει καμία. Η εκπροσώπηση λοιπόν των γυναικών στα ε, διοικητικά συμβούλια και προβάλλονται δύο βασικά επιχειρήματα. Καταρχάς έχουμε το επιχείρημα της περισσότερης δικαιοσύνης και περισσότερης ισότητας, αλλά υπάρχει και το οικονομικό σκέλος, δηλαδή ένα επιχείρημα υπέρ της οικονομικής δραστηριότητας. Από την ηθική σκοπιά του θέματος είναι προφανές ότι η γυναίκα πρέπει να εκπροσωπείται επί ίσης όρης συγκριτικά με τους άντρες στα ΔΣ. Άλλωστε, οι γυναίκες είναι ε, πάνω από το 50% των φοιτητών στα πανεπιστήμια και των πτυχιούχων τελικά. Προβάλλεται το επιχείρημα ότι εάν υπάρξουν περισσότερες γυναίκες στα, διπλω... στα διοικητικά συμβούλια, αυτό θα αποτελέσει καθρέφτη και καταλήτη ώστε να αυξηθούν και οι γυναίκες στο middle management, στα μεσαία ε, διοικητικά στελέχη. Και ορισμένες μελέτες ε, υποδεικνύουν ότι πράγματι υπάρχει αυτή η σχέση, αυτός ο συσχετισμός θα έλεγα ότι είναι περισσότερο συσχετισμός και όχι τόσο σχέση αιτίου αιτιατού. Δεν είναι το ίδιο αυτά τα δύο. Ως προς το οικονομικό επιχείρημα που έχει προβληθεί, το είπαν και οι προηγούμενες ομιλήτρες, η μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών στα ΔΣ αυξάνει την αξία της επιχείρησης και άρα αυξάνει την απόδοσή της, τα έσοδά της, την οικονομική της αξία. Και από αυτή την πλευρά διάφορα προ... επιχειρήματα προβάλλονται. Η παρουσία των γυναικών αυξάνει την ανεξαρτησία των διοικητικών συμβουλίων, προσφέρει νέες γνώσεις, νέες οπτικές γωνίες, εντείνει τη δημιουργικότητα, εκδίδονται και στέλνονται θετικά μηνύματα στις αγορές ε, ε, εντείνεται η δραστηριότητα της επιχειρήσης, υπάρχουν διαφορετικά στυλ και τρόποι ηγεσίας, κάτι το οποίο εμπλουτίζει την ε, ηγετική δραστηριότητα αλλά και τη διοίκηση γενικότερα. Και σύν τις άλλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες ε, παρίστανται περισσότερο, είναι περισσότερο παρούσες στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων συγκριτικά με τους άνδρες. Ωστόσο, άλλες μελέτες τείνουν να ε, καταδεικνύουν ότι η παρουσία των γυναικών ενδεχομένως θα ήταν ερνητική για την αξία της επιχείρησης. Και τι επικαλούνται όσοι το ε, υποστηρίζουν. Λένε ότι δεν θα είναι ομοιογενής η ομάδα στο διοικητικό συμβούλιο, Επομένως, κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης θα χρειαστεί περισσότερο χρόνος, περισσότερο χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί και προβάλλουν το εξή επιχείρημα, ότι οι γυναίκες δεν είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων λόγω των δικών τους επαγγελματικών χαρακτηριστικών. Άρα η παρουσία τους μπορεί να ε, θεωρηθεί αρνητική και να αποβεί αρνητική για την αξία της επιχείρησης. Αυτό το επιχείρημα προβάλλεται, με το οποίο βεβαίως εγώ διαφωνώ. Όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι είναι σημαντική και θετική η σχέση μεταξύ της παρουσίας των γυναικών στα ΔΣ και της αξίας της επιχείρησης αυτής κάθε αυτής. Και σε αυτό το πίδακα βλέπουμε τις διάφορες μελέτες που έχουν εκπονηθεί. Είναι αληθές ότι οι πρώτες μελέτες που ε, εκπονήθηκαν σε γενικές γραμμές έδειχναν ένα θετικό απολογισμό, ένα θετικό ισοζύγιο. Όμως ε, δεν έλαβαν υπόψη τους διάφορα θέματα. Μία μελέτη δείχνει ότι ο συσχετισμός είναι αρνητικός και άλλες μελέτες δείχνουν ότι ο συσχετισμός είναι ουδέτερος. Δηλαδή ότι η μεγαλύτερη προσώπηση γυναικών στα ΔΣ τελικά δεν έχει ούτε αρνητικό ούτε θετικό αντίκτυπο στην αξία της επιχείρησης. Γιατί λοιπόν έχουμε μελέτες με διαφορετικά πορίσματα. Πρώτον διότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στην έρευνα. Σχεδιάζεται διαφορετικά η εκάστοτε μελέτη, τα δείγματα είναι διαφορετικά, η χρονική περίοδος δειγματοληψίας είναι διαφορετική, η επιλογή των χωρών είναι διαφορετική. Επίσης, η διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων καθορίζεται και ε, η επίπτωση του φύλου στις επιδόσεις, στην απόδοση ε, είναι κάτι που αξιολογείται διαφορετικά και τελικά αυτό το οποίο προκύπτει είναι ένας συσχετισμός. Δηλαδή όσο περισσότερες γυναίκες στο ΔΣ τόσο μεγαλύτερη αξία της επιχείρησης. Αυτό όμως είναι άλλο και άλλο η... το αιτιατό. Δηλαδή μπορεί οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη αξία να είναι αυτές που θέλησαν και απέκτησαν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά του συμβούλια. Δεν είναι απαραίτητο ότι η παρουσία των γυναικών είναι αυτή που αύξησε τη τιμή ως αποτέλεσμα. Είναι πιθανό δηλαδή ε, τελικά να μην υπάρχει σχέση βάσει συγκεκριμένων μελετών. Και είναι λογικό αυτό, γιατί ακόμα και οι μελέτες που πιστεύουν ότι υπάρχει σχέση αιτίου αιτιατού δεν θεωρούν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ π.χ. της παρουσίας ανεξάρτητων συμβούλων στην επιχείρηση και της αξίας αυτής καθεαυτής της επιχείρησης. Άλλο πράγμα δηλαδή ο συσχετισμός τελικά, υπάρχει συσχετισμός και άλλο πράγμα το ότι το ένα προκαλεί και είναι γενεσιουργός αιτία του άλλου. Από επιστημονική σκοπιά ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντοτε η σχέση είναι θετική και στατιστικό σημαντική. Άλλωστε αυτό είναι ένα πείραμα που μπορούμε να κάνουμε στην, ε, ε, κατά τη θέσπιση του κώδικα δεοντολογίας αλλά και των ποσοστώσεων σε ορισμένες χώρες γίνεται ανάλυση των ε, πειραματισμών των φυσικών αν θέλετε. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε μελέτες που έχουν δείξει ότι ορισμένες επιχειρήσεις επωφελούνται περισσότερο από αυτή τη διαφοροποίηση των φύλων από ότι άλλες επιχειρήσεις. Ενώ άλλες επιχειρήσεις ε, βλέπουμε ότι άπαξ και λάβουν υπόψη τα χαρακτηριστικά ε, γυναικών και ανδρών, δηλαδή την ηλικία τους και την επαγγελματική τους κατάρτιση και δεξιότητες, τελικά δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές για άλλες επιχειρήσεις. Ε, στατιστικό σημαντικές διαφορές ε, που να συσχετίζουν την παρουσία γυναικών με την αύξηση της αξίας της επιχείρησης. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πραγματικά ωφέλη συνδέονται με την προσέλκυση στα ΔΣ γυναικών που έχουν γνώσεις που έχουν σχέση με την επιχείρηση. Και τι συμβαίνει τώρα με τις ποσοστώσεις. Έχουμε κάποια στοιχεία για την ε, ε, θετική επίπτωση των ποσοστώσεων. Είναι πρόσφατες οι μελέτες αυτές, δεν έχουμε πάρα πολλά ε, στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, οι μελέτες δείχνουν ότι οι ποσοστώσεις ήταν πολύ αποτελεσματικές, π.χ για την αύξηση των γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια αλλά όχι σε επίπεδο μεσαίας και υψηλής διοίκησης. Δηλαδή είναι αποτελεσματικό να έχουμε περισσότερες γυναίκες ως μέλη διοικητικών συμβουλίων, αλλά αυτό δεν οδηγεί στην πρόσληψη περισσότερων γυναικών στις εκτελεστικές θέσεις και γενικότερα στη διοίκηση, ε, ε, τη διοικητική ιεραρχία αυτής της επιχείρησης. Και σύν της άλλης υπήρξε πρόβλημα με την εφαρμογή των ποσοστώσεων, γιατί αν δεν έχουμε αρκετές γυναίκες σε εκτελεστικές και επιτελικές θέσεις, τότε είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό γυναικών που θα μπορούσε να στελεχώσει ε, τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Στον πανεπιστημιακό κύκλο αυτό μπορεί να συμβεί. Σε πολλές χώρες το ποσοστό γυναικών που είναι τακτικές ε, καθηγήτριες, ε, έχουν τη θέση δηλαδή του τακτικού καθηγητή, έχει αυξηθεί 20%. Αυτό το βλέπουμε και στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Τούτων λεχθέντων εμείς, οι γυναίκες, ε, έχουμε πολλά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουμε για να φτάσουμε στις ανώτατες επιτελικές θέσεις των επιχειρήσεων. Όχι όμως μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και των κυβερνήσεων. Δείτε τη σύνθεση των κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο σε επίπεδο υπουργών, αλλά και πιο κάτω. Υφυπουργών και το καθεξής. Και εκεί βλέπουμε ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται. Το ίδιο συμβαίνει και στα συνδικάτα. Το ίδιο συμβαίνει στα νοσοκομεία, όπου αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες το 50% των γιατρών είναι γυναίκες, αλλά διευθυντές κλινικής είναι το 10% γυναίκες ή και στον τομέα των θετικών επιστημών ή των επιστημών γενικότερα. Ε, τακτική, τακτικές καθηγήτριες είναι το 10-20% και αν δούμε πόσοι πρίτανεις είναι γυναίκες στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ε, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ λίγες και ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται για τις ε, θέσεις των πριτάνων και το καθεξής. Το ίδιο βέβαια ισχύει και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με χαμηλή παρουσία γυναικών στις ε, υψηλές θέσεις. Τούτο λεχθέντων. Το συμπέρασμα είναι ότι τα εμπειρικά στοιχεία δεν μας παρουσιάζουν ξεκάθαρα ως συμπέρασμα το ότι αυξάνει η αξία της επιχείρησης με την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα ΔΣ. Αυτό το επιχείρημα δεν είναι πολύ σαφές. Θα πρέπει να βασαστούμε στα επιχειρήματα της ηθικής και της δικαιοσύνης. Εγώ προφανώς πιστεύω ότι τα εμπόδια και οι φραγμοί θα πρέπει να αρθούν και να καταρριφθούν. Βεβαίως πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Αυτό που δείχνουν μάλλον οι ποσοστώσεις είναι ότι δεν έχουν αντίκτυπο στα, στους άλλους τομείς της επιχείρησης, στη διοίκησή της και μάλιστα μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα και είναι ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό, αναπάντητο. Δηλαδή, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ένας μέτοχος ε, διακινδυνεύει τα χρήματά του και περιμένει να έχει αντίστοιχη απόδοση ε, αναλόγως με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εάν θεσπίσουμε κάτι τέτοιο και δεν το θεσπίσουμε π.χ. στα δημόσια πανεπιστήμια, δεν το θεσπίσουμε στις κυβερνητικές θέσεις ή και σε άλλους τομείς της δημόσιας σφαίρας, ουσιαστικά η άποψή μου η προσωπική είναι ότι θα, ε, δεν θα, ε, θα είναι σαν να μην ε, μεταχειριζόμαστε ευνοϊκά τις επιχειρήσεις και να μεταχειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο τις κυβερνήσεις και τους άλλους τομείς της δημόσιας σφαίρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. κυρία Γκόμες Ανσόν για την ε, συμβολή σας ε, στο εργαστήρι μας. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τους άλλους εμπειρογνώμενες στο Προεδρείο για να... Μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η κυρία Ζούμπια Χόκροφτ είναι η επόμενη ομιλήτρια η οποία ε, είναι εμπειρογνώμη στο θέμα των ε, προσλήψεων υψηλόβαθμων στελεχών σε μη, εκτελε, σε μη εκτελεστικές ε, διευθυντικές θέσεις στην Ευρώπη του γραφείου MSC Headhunters. Καλό σας απόγευμα. Είμαι η Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία MSC Headhunters, δηλαδή μια εταιρεία κυνηγών επιχειρηματικών στελεχών ε, και επίσης ε, συμμετέχει στο πάνελ ε, αυτό και η παρουσίασή μου βασίζεται και στη συμμετοχή στελεχών του Πανεπιστήμιου του Μάντσεστερ. Θα σας εξηγήσω ε, πώς λειτουργεί η διαδικασία πρόσληψης υψηλόβασμων στελεχών, το ιστορικό της διαδικασίας αυτής και γιατί ε, πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, γιατί είναι επίκαιρα και σχετικά με το θέμα που συζητάμε γενικώ και γιατί, τι εμπόδια, τι προσκόμματα υπάρχουν ε, που, για τις γυναίκες να συμμετάσχουν ε, σε εκτελεστικές θέσεις και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να ξαναπεράσουμε αυτά τα εμπόδια.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 Ε, ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα να χρησιμοποιούμε μια τέτοια διαδικασία, ένα τέτοιο στελεχός για να βρει τα διοικητικά στελέχη είναι ότι είναι πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική. Επίσης στοχεύει συγκεκριμένα σε προσόντα και δεξιότητες και ο ρόλος μας είναι να ε, εκπαιδεύσουμε και να ενημερώσουμε τα άτομα αυτά για τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να προσεγγίσουμε και να ταυτοποιήσουμε αυτά τα άτομα παρά μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας. Λοιπόν, δεδομένου ότι οι θέσεις αυτές είναι πολύ ειδικέ και πολύ συγκεκριμένε, εμείς προσπαθούμε να ταιριάξουμε τις ανάγκες ε, την προσφορά με τη ζήτηση. Και επίσης ε, το ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι όλοι μας οι υποψήφοι καλύπτονται από την αρχή της εμπιστευτικότητα, διότι όλες οι θέσεις μας είναι top secret, είναι εξαιρετικά εμπιστευτικέ έτσι ώστε να μην διαρρεύσουν πληροφορίες στους ανταγωνιστές ε, της επιχείρησης και γενικά στην αγορά. Υπάρχουν ε, λοιπόν μοναδικές ε, προσεγγίσεις, μοναδικές οπτικές γωνίες σε αυτό, το, τη δεξιότητα, σε αυτό το στέλεχος που προσπαθεί να ενορπίσει άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Ανοίγει ένα παράθυρο λοιπόν αυτό το στέλεχος σε δύο ε, τομείς. Πρώτον, στους ε, πελάτες μας από πλευράς επιχειρηματικού κόσμου και δεύτερον, στους υποψήφιους. Ε, ενημερώνουμε ε, τους υποψήφιους πολύ συγκεκριμένα για την περιγραφή του, της εργασίας τους, τις προδιαγραφές ε, της θέσης, συζητούμε τα προσωπικά τους δεδομένα, τις φιλοδοξίες τους για καριέρα, τις τα εικονιακά τους δεδομένα Δηλαδή ε, όλες τις ε, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές ε, γωνίες και προσεγγίσεις τις συζητούμε με τους υποψήφιους. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, εάν ανοιχτεί μια θέση, παρουσιαστεί μια θέση στην αγορά, υπάρχει δηλαδή ζήτηση για μια θέση, θα προσεγγίσουμε περίπου 100 100 υψηλόβασμα στελέχη για αυτή τη θέση. Μιλάμε λοιπόν για μια πάρα πολύ ενδελυχή και εις βάθος εξέταση όλων των ε, δεξιοτήτων προσόντων του υποψήφιου για να, τον, να δούμε αν ταιριάζει σε αυτή τη θέση. Η στόχη μας λοιπόν είναι να κατανοήσουμε τα προσκόμματα που υπάρχουν όσον αφορά την πρόσληψη γυναικών και τις συστάσεις που μπορούμε να υλοποιήσουμε για την εξάλληψη αυτών των προσκομμάτων. Τώρα, όταν μιλάμε για, διάκριση, διακρίσεις που βασίζονται στο φύλλο, ή όπως εγώ προτιμώ, αντί για discrimination να πούμε differences, διαφορές ε, φύλου. Ε, αυτό που θέλουμε να καταρχάς ε, να, πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι υπάρχουν αρνητικές αντιλήψεις όσον αφορά τις γυναίκες. Πολλοί λένε ότι οι γυναίκες δεν θέλουν αυτές τις ε, θέσεις. Έχουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν αυτές αυτό το επίπεδο καθηκόντων και υποχρέωσεων ίσως όπως πρέπει να συμπεριφερθούν ακριβώς όπως οι άντρες όταν ανεβούν ε, στην, στα δικαιωτικά συμβούλια, στην καριέρα τους. Ε, γι' αυτό ακριβώς οι δεξιότητες και τα προσόντα είναι πολύ πιο σημαντικά από τις πολιτιστικές ε, από τα πολιτιστικά στοιχεία. Πολλές φορές λοιπόν επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στη διαδικασία πρόσληψης, στην καταλληλότητα. Αν είναι κατάλληλο το άτομο αυτό, αν έχει την εμπειρία, και όχι μόνο τις ε, ικανότητες. Επίσης, ε, πολλές φορές οι γυναίκες δεν αισθάνονται άζεντα, θυματοποιούνται μέσα σε ένα αποκλειστικά αντρικό περιβάλλον, η οργανωτική δομή της επιχείρησης δεν έχει διαφάνεια, οι άντρες δεσπόζουν και έτσι οι γυναίκες δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση, ε, ιδίως όταν θέλουν να συνεργαστούν με άλλες γυναίκες. Βλέπετε ότι πολλές φορές οι γυναικείες θέσεις ε, τις καταλαμβάνουν <clears throat> στις διευθύνσεις προσωπικού, δημοσίων, σχέσεων και παρόμοια δηλαδή ε, διευθύνσεις μέσα στις επιχείρησεις και δεν ανεβαίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν προβιβάζονται. Πιστεύω λοιπόν ότι η πιο το πιο κρίσιμο σημείο, το κέριο σημείο που είναι εμπόδιο για την άνοδο των γυναικών είναι αυτή ακριβώς η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ της κονιακής ζωής και του εργασιακού βάρους. Δηλαδή δεν υπάρχει ε, τη δυνατότητα να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. Υπάρχουν ατελείωτες ώρες εργασίας, έλλειψη ευελιξίας, το ξέρω κι εγώ προσωπικά. Ε, δεν... Ε, πολλές επιχειρήσεις πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να παρέχουν ορισμένες διευκολύνσεις στις ε, γυναίκες για να μπορούν να μοιραστούν ακριβώς αυτό το κοινιακό βάρος μεταξύ στελέχους και μητέρας. Ε, δεν υπάρχει πολλές φορές και η στήριξη από την, ε, πιο, την προηγούμενη γενιά, δηλαδή τους πιο μεγάλους σε ηλικία. Όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών, οι εταιρείε δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό θα, θα πρέπει να παρέχουν έχετε μέσα στην επιχείρηση, εντός της επιχείρησης, διότι είναι εξαιρετικά μεγάλο το κόστος ενός νηπιαγωγείου, ενός παιδικού σταθμού. Έχω δει λοιπόν διαπιστώσει σε πολλές περιπτώσεις όταν μια εταιρεία θέλει να προσλάβει ψηλόβαθμο στέλεχος ότι οι μητέρες δεν θεωρούνται επιλέξιμες. Αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό, καταλαβαίνετε, για μια γυναίκα που έχει παιδιά να απορρίπτεται με αυτό το κριτήριο. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να συμβαδίσει η δουλειά με τη μητρότητα. Τώρα, ε, τι μπορεί να αλλάξει οι συστάσεις μας θα έλεγα ότι να ξεκινήσουμε με την ε, συνειδητοποίηση και την εκπαίδευση του προβλήματος. Θα πρέπει οι γυναίκες να ε, τις στηρίξουμε όσον αφορά την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους, ε, την ενίσχυση του εγώ τους, του πιστεύω τους, να πιστέψουν ότι μπορούν να αναλάβουν αυτούς τους ρόλους. Ο η διευθύνουσα σύμβουλος του Facebook έχει γράψει πρόσφατα ένα βιβλίο όπου λέει ότι οι γυναίκες θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβουν περισσότερες ε, θέσεις υψηλόβαθμες και στα διοικητικά συμβούλια και θα πρέπει να διευκολύνουμε τις γυναίκες να γίνουν πιο φιλόδεξες εφόσον το επισημούν. Είναι πάρα πολύ λίγες οι θέσεις που υπάρχουν για αυτές και γενικά το... είναι πάρα πολύ ωφέλιμη η συμμετοχή τους. Τώρα, τι θα πρέπει να κάνουν οι εταιρείε. Θα πρέπει να υποβάλουν ένα, μια ετήσια έκθεση για την σύνθεση του φύλου στα διοικητικά του συμβούλια, ε, να δεσμευθούν όσον αφορά την ισότητα του φύλου και εάν δείτε τις εισηγμένες εταιρείε στο Βρετανικό χρηματιστήριο Υπάρχουν μόνο 7 διοικητικά συμβούλια συγμένων εταιριών που έχουν μόνο άνδρες στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν αλλάζει η κατάσταση σιγά σιγά. Και όσον το αφορά τώρα τα κριτήρια προσλήψεων, θα πρέπει να υπάρχει ένας εθελοντικός κώδικας ε, συμμόρφωσης και της εφαρμογή, να δημοσιεύονται ε, τα μη εμπιστευτικά, ε, οι μη εμπιστευτικές θέσεις και απόψεις των συμβουλίων, να αυξηθεί η εστίαση στις δεξιότητες, να επιλέγονται ε, όχι μόνο ε, να μην υπάρχει μόνο διάκριση του φίλου ε, αλλά να διαλέγουμε πάντοτε τον καλύτερο τον καλύτερο άντρα, την καλύτερη γυναίκα βέλτιστη επιλογή θα ήθελα λοιπόν να, να δούμε πού διαφωνούμε και θα ήθελα να σας προσθέσω τώρα λίγο, ε, να σας κάνω μια κάπως πρόκληση με την παρουσίασή μου αυτή για το πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το χάζα μεταξύ των δύο φίλων και να γίνουν περισσότερες γυναίκες ε, μοντέλα στο ρόλο τους. Ε, είχα λοιπόν ορισμένες διαφωνίες με τους συναδέλφους μου ε, για τη δική μου προσέγγιση και δεδομένου ότι μπορώ να σας μιλήσω από τη δική μου θέση και από τη δική μου εμπειρία πρέπει να πω ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο φιλόδοξες μόνο 5% σε όλες τις έρευνες που κάναμε ε, ήταν γυναίκες υποψήφιες, δηλαδή δεξαμενή υψηλόβασμων στελεχών από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε υποψήφιες ή υποψήφιους είναι πάρα πολύ μικρή για τις γυναίκες, μόνο 5% οι γυναίκες θέλουν να δίνουν την εντύπωση ότι είναι πιστές στον εργοδότη τους, ε, έχουν μειωμένες φιλοδοξίες και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αυτοπεποίθηση ε, και το πρόβλημα το μεγάλο βεβαίως το οικογενειακό. Ε, γι' αυτό ακριβώς από τη δική μας προοπτική τα επιπτώσεις είναι αρνητικές στις γυναίκες ε, λόγω αυτού υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στον ε, τομέα και πολλές φορές προσλαμβάνονται λανθασμένα άτομα για, την, για τη θέση. Λανθασμένοι υποψήφοι. Και ε, έτσι δημιουργούνται και αρνητικές προσεγγίσεις, μια αρνητική αντίληψη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, υπάρχει αυτό το δεδομένο. Δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες που να μπορέσουν μέχρι το 2020 να πληρώσουν αυτές ε, τις ποσοστώσεις που έχουν οριστεί και γι' αυτό οι προσπάθειές μας πρέπει να γίνουν πιο έντονες και η κατάσταση είναι κρίσιμη. Πρέπει να ενισχύσουμε τις γυναίκες, να τους δώσουμε τα μέσα εκείνα τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να περνάνε μέσα από το σύστημα και να καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις. Ευχαριστώ που μας μίλησατε για την εμπειρία σας ε, από τον τομέα των προσλήψεων και τις πρακτικές που υπάρχουν. Πάμε στον επόμενο ομιλητή, Kim Peters, που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου του Exeter για τα ψυχολογικά στοιχεία και οικονομικά στοιχεία που διέπουν τη συμμετοχή των γυναικών σε επιτελικές θέσεις. Πριν δώσω το λόγο Θέλω να σας πω ότι όλες τις ομιλίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε online και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν μπορείτε να δείτε αυτές τις παρουσιάσεις και αργότερα. Κυρία Πίτερ, έχετε τον λόγο. Είσαστε στα αριστερά μου. Πάντα στα αριστερά μου οι ομιλίτες, Βλέπω. Με μεγάλη χαρά άκουσα τη Ζούμπια, γιατί μίλησε πραγματικά από την εμπειρία σας, ε, την εμπειρία της, ε, για το πώς ε, προσεγγίζουν τις ηγετικές θέσεις οι γυναίκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την έρευνα που κάναμε εμείς σε ό,τι αφορά την ψυχολογία των γυναικών σε αυτές τις θέσεις, στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ. Ξέρετε πολύ καλά ότι υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες, όχι μόνο στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, αλλά και σε όλες τις υψηλέ και σημαντικέ θέσει. Η εξήγηση. Γιατί συμβαίνει αυτό. Οι εξηγήσει την τελευταία δεκαετία άλλαξαν πολύ. Αν κοιτάξετε δηλαδή το 1980, τότε εστιάζαμε στα, στους φραγμούς που αντιμετώπισαν οι γυναίκες. Ε, τότε μιλούσαμε για το γυάλινο, α, τη γυάλινη οροφή. Δηλαδή, φτάνανε μέχρι τις μεσαίες επιτελικές θέσεις και μετά δεν μπορούσαν να σπάσουν αυτό το όριο, ας πούμε. Ε, υπήρχαν τότε και διακρίσεις Λέγαν τότε, α πούμε, ότι οι γυναίκε δεν είναι τόσο καλέ όσο οι άντρες εκείνη την εποχή, αλλά άλλαξαν τα πράγματα. Αν τώρα στη Δύση ρωτήσεις ε, η ικανότητα των γυναικών είναι επαρκή. δεν θα ακούσει τι ίδιε προκαταλήψεις που άκουγε παλιά. Επίσης, ε, τα εμπόδια δεν είναι απαράλλαχτα και αναλύωτα. Μερικέ φορές σπάνε αυτή την ε, γυάλινη οροφή οι και φτάνουν στι ανώτατε θέσει. Προσπαθήσαμε τώρα να, εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει και βλέπουμε ότι αν κάποιες γυναίκες τα καταφέρνουν, τίθεται ερώτημα γιατί δεν μπορούν να τα καταφέρουν περισσότερες. Τότε οι περισσότεροι δίνουν την απάντηση ότι οι γυναίκες απλώς δεν θέλουν. Ε, δεν έχουν την ε, φιλοδοξία. Δηλαδή ε, προτιμούν την ισορροπημένη ζωή, θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, προτιμούν να μην σκαρφαλώσουν ψηλά στην ιεραρχία. Αν κοιτάξετε την, τη βιβλιογραφία υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι δείχνουν μικρότερη φιλοδοξία για την καριέρα τους από τους άντρες. Εμείς το, στην έρευνα που κάναμε στο Πανεπιστήμιο του Exeter ε, προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι αυτή η παρατήρηση ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο φιλόδοξες ε, δεν οφείλεται στο ότι από τη φύση τους είναι λιγότερο φιλόδοξη, ότι υπάρχει μια βιολογική διαφορά, ας πούμε, μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τη φιλοδοξία. Απλώς έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Μπαίνουν, ας πούμε, στις εταιρείε με την ίδια φιλοδοξία ε, οι γυναίκες, αλλά η ίδια η οργάνωση, οι ίδιες οι εταιρείες, η ίδια η κουλτούρα που υπάρχει διαβρώνει αυτή τη φιλοδοξία. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν πώς αφομοιώνουν αυτή την εμπειρία οι γυναίκες. Και θα συζητήσω ε, τρία διαφορετικά, τρεις διαφορετικές έρευνες ε, που κάναμε για να καταλάβουμε την ψυχολογία των γυναικών και για το τι υποσκάπτει η φιλοδοξία τους. Θα μιλήσω λοιπόν για τη σημασία των της αντίληψης των εργοδοτών τους. Οι γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις ε, δεν πιστεύουν ότι είναι κατάλληλες για να ηγηθούν. Επίσης υπάρχει ο λεγόμενος γυάλινος ε, γκρεμός. Ε, μερικές φορές, αυτό, ο οποίος περιγράφει το είδος των ηγετικών θέσεων που καταλαμβάνουν οι, θέσεις, οι γυναίκες. Δηλαδή έχουν την τάση να τους δίνουν πιο αβέβαιες, πιο σταθείς ηγετικές θέσεις. Και επίσης αμείβονται λιγότερο οι γυναίκες από τους άντρες στις ίδιες θέσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία ε, διαβρώνουν τα κίνητρά τους και τη φιλοδοξία τους. Πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, πάμε να δούμε τις αντιλήψεις. Και από την έρευνά μας προκύπτει ότι σε περισσότερες εταιρείε και οργανώσεις, άντρες και γυναίκες που πιστεύουν ότι είναι διαφορετικοί από αυτούς που πέτυχαν, εκείνοι οι ίδιοι δεν αισθάνονται ικανοί να πετύχουν. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ ε, πώς ε, βλέπεις τον εαυτό σου, ε, πώς φαντάζεσαι ότι θα προχωρήσεις, μπορείς να τα καταφέρεις, κοιτάς γύρω σου. αν πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, τότε υπάρχουν περισσότερα ποσοστά επιτυχίας. οι άνδρες και οι γυναίκες βλέπουν διαφορετικά τον εαυτό τους. Ε, γιατί να κάνεις θυσίε ε, αν δεν πιστεύεις ήδη από την αρχή ότι θα τα καταφέρεις. Στους περισσότερους τομείς υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα στην ε, θέση του διευθυντή και στο φίλο του άντρα. Όταν οι άντρες, λοιπόν, όταν οι γυναίκες βλέπουν το μέλλον τους, βλέπουν ότι τη διευθυντική θέση θα την καταλάβει ένας άντρας. Ενώ όταν ε, ένα άντρα κοιτάζει γύρω του, α πούμε, τι συμβαίνει, κοιτάζει του μεγαλύτερου του, σε τι θέσει είναι κτλ., βλέπει στι διευθυντικέ θέσει ότι υπάρχουν άντρε. Υπάρχει αυτή η ταύτιση. Σε πολλά επαγγέλματα βλέπουμε ότι οι γυναίκε βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πολλέ γυναίκε ε, σε ηγετικέ θέσει. Αυτό μειώνει τα κίνητρά του να προσπαθήσουν να καταλάβουν τέτοιε θέσει. Η δεύτερη έρευνά μα είναι να δούμε τι συμβαίνει όταν καταφέρουν οι γυναίκες να σπάσουν αυτή την ε, γυάλινη οροφή και να πετύχουν την ε, επιτελική θέση. Τι δείχνει η έρευνα. Ότι οι γυναίκες κατά πάσα πιθανότητα θα διοριστούν σε επικίνδυνες ηγετικές θέσεις, οι επιτελικές θέσεις. Σε πολλές ε, έρευνες ρωτήσαμε ανθρώπους να υποδείξουν, ας πούμε, ποιος θεωρούν ότι είναι ο κατάλληλος για μια διευθυντική θέση ένας ένα πούμε, και μία γυναίκα. Όταν ε, θέλουν, ε, όταν πρόκειται να διορίσουμε έναν διευθυντή σε μια επιτυχημένη εταιρεία, οι περισσότεροι έχουν την τάση να προτιμούν έναν άντρα. Ενώ όταν ε, πρόκειται να διορίσουμε μια, ένα διευθυντή σε μια αποτυχημένη εταιρεία, η τάση να διορίσουμε μια γυναίκα. Υπάρχουν δηλαδή στερεότυπα. Υπάρχουν βέβαια και θετικά στερεότυπα υπέρ των γυναικών αλλά και αρνητικά. Μερικέ φορές, α πούμε, λέμε ότι είναι καλέ στην επικοινωνία οι γυναίκε. αλλά συχνά ταυτίζουμε την κρίση με το γυναικείο φύλλο. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Δίνουμε ευκαιρίε για ηγετικέ θέσει στι γυναίκε, αλλά αυτέ οι ευκαιρίε δεν είναι ακριβώ οι ίδιε ευκαιρίε με τι ευκαιρίε που έχουν οι άντρε. Είναι πολύ πιο αγχωτικέ, έχουν υψηλότερο ρίσκο αποτυχία. Οι επιπτώσει για τι γυναίκε ποιε είναι, ότι αυτή η αγχωτική εμπειρία δεν δίνει κίνητρα και μειώνει την επιθυμία σου να προχωρήσει, αντίθετα αυξάνει την επιθυμία σου να τα παρατήσει. Η τρίτη έρευνα αφορά το, τη διαφορετική αμοιβή άνδρων και γυναικών. Το ξέρετε αυτό το φαινόμενο όλοι. Οι γυναίκε, δηλαδή πληρώνται λιγότερο από τους άνδρες για να κάνουν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Αυτό το κενό των αμοιβών ε, αυξάνεται όσο ανεβαίνει στην ιεραρχία. Η έρευνα μας δείχνει ότι ένας από τους λόγους γι' αυτό είναι πάλι τα στερεότυπα που έχουμε για τις γυναίκες και τους άντρες. Δηλαδή, υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται ο, τι πιστεύουμε για την ηγετική θέση. Ε, κοιτάμε, ας πούμε, το πώς θα πάει μια εταιρεία και πιστεύουμε ότι όταν, ας πούμε, επιτυγχάνει, ε, οφείλεται στο διευθυντή, όταν αποτυγχάνει πάλι οφείλεται στον, ε, στο διευθυντή. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τα υπόλοιπα στοιχεία. Η έρευνα μας δείχνει ότι αυτό το, αυτή την τάση την, ε, και αυτή την ε, σκέψη την εφαρμόζουμε πολύ περισσότερο στις γυναίκες. Δηλαδή αν αποτύχει μια εταιρεία θεωρούμε ότι φταίει η γυναίκα. Ε, η γυναίκα είναι πιο ανίκανη να τα καταφέρει σε μια ηγετική θέση αλλά μπορεί να βοηθήσει, είναι καλή στην επικοινωνία κτλ. Ε, δηλαδή, οι άντρες τελικά ε, αμείβονται για την επιτυχία μιας εταιρεία, ενώ οι γυναίκες όχι. Επομένως αυτό έμεσα τι σημαίνει ότι η προσπάθειά σου δεν αξίζει τόσο πολύ, πολύ όσο οι προσπάθειες των ανδρών. Και άρα δεν πρέπει να σε να αμύψουμε το, το ίδιο. Αυτό τι σημαίνει ότι αυξάνει η επιθυμία σου πάλι να τα παρατήσεις και αντίθετα μειώνει την επιθυμία σου να προχωρήσεις. Η έρευνα μας δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές στις ε, φιλοδοξίες καριέρας ανδρών και γυναικών, αλλά όχι γιατί οι γυναίκες από τη βιολογία τους, από το λόγο φίλου, είναι λιγότερο φιλόδοξες. Αυτό οφείλεται στην εμπειρία που, που ζουν, στις εμπειρίες που ζουν, ε, μπαίνοντας σε μια εταιρεία, σε μια οργάνωση κτλ. Ε, οι γυναίκες κοιτάνε γύρω τους, δεν βλέπουν αρκετούς επιτυχημένους ανθρώπους σαν κι αυτές, δηλαδή γυναίκες. Επίσης, δεν αμείβονται για την επιτυχία τους με τον τρόπο που αμείβονται οι άντρε. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Αν θέλετε να βοηθήσετε τις γυναίκες να ανέβουν πιο ψηλά σε μια οργάνωση, σε μια εταιρεία, θα πρέπει να σκεφτείτε την ψυχολογία τους που δημιουργήθηκε λόγω εμπειρίας και τι τις κινητοποιεί και αντίθετα τι δημιουργεί αντικίνητρα για την εξέλιξή τους. Σας ευχαριστώ πολύ και τη συνεισφορά σας στη συζήτηση. Τώρα θα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Χάχα. Ένα λεπτό μόνο. Έτσι είχαμε σκεφτεί τουλάχιστον. Να δώσω σε αυτό το σημείο την ευκαιρία στα μέλη της Επιτροπής μας να πάρουν το λόγο. Η κυρία Ρέγνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση προς την κυρία Hawthorne, μια ρεαλιστική ερώτηση όσον αφορά τα κριτήρια προσλήψεων. Όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη διαδικασία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, αδιάβλητα αντικειμενικά κριτήρια όσον αφορά την αξιολόγηση των σπουδών, των διπλωμάτων, των πτυχίων κλπ. Ε, υπάρχουν λοιπόν και υποκειμενικά, υποκειμενικά κριτήρια ε, τα οποία λένε ότι πρέπει ο υποψήφιος να έχει, να είναι δυναμικός χαρακτήρας, να δείχνει ευελιξία, διάθεση συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα κλπ. Ποια είναι οι εμπειρία σας λοιπόν όσον αφορά αυτά τα υποκειμενικά κριτήρια έναντι των αντικειμενικών. Και αυτό που είπατε ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο φιλόδοξες. Μήπως αυτό έχει σχέση με τα στερεότυπα αυτά τα οποία ακριβώς σχετίζονται με τα υποκειμενικά κριτήρια. Ευχαριστώ, ε, κυρία Κόχενρη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Μία προς την κυρία Χόκροφτ. Όταν μιλήσατε για τις εκτελεστικές θέσεις είπατε ότι 100 ε, ενδυνάμει είναι υποψήφοι για μία θέση. Πόσες ε, εκ των 100 είναι οι γυναίκες. Π.χ. 50 γυναίκες και 50 οι άνδρες μπορούν να ε, διεκδικήσουν δικαίως τη θέση αυτή. Αυτή είναι η πρώτη... Να το απαντήσω τώρα. Προσπάθησα να το εξηγήσω. Όχι, συγγνώμη, τη διακόπτει ο πρόεδρο. Θα ακούσουμε όλε τι ερωτήσει μαζί και μετά θα μπορέσετε να απαντήσετε όταν σα δοθεί ο λόγο. Επόμενο ερώτημά μου λέει η βουλευτή είναι το εξή. Όταν μιλούμε για την ευελιξία και αν δούμε την προσωπική ζωή ενός υποψηφίου ή μίας υποψήφιες, υποψήφιες. Το συζητάτε αυτό με έναν άνδρα. Π.χ. τον ρωτάτε πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να πάρεις τα παιδιά σου από το σχολείο. Ε, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό όταν έχετε άνδρα υποψήφιο στο κυνήγι κεφαλών που κάνετε. Ε, εγώ έχω την εξή εμπειρία. Οι γυναίκες που είναι σε ηγετικές θέσεις μιλούν γι' αυτό από μόνες τους και οι άνδρες δεν μιλούν ποτέ γι' αυτό, εκτός και αν τους ρωτήσει κανείς ποιο μερίδιο ευθύνης στην, στην οικογενειακή ζωή αναλαμβάνεται και πόσο μερίδιο ευθύνης αφήνεται στις συζύχους σας. Είναι αυτό μέλος, μέρος της τεχνικής της ε, συνέντευξης. Δεν το λέω για να σας επικρίνω, απλά με ενδιαφέρει να μάθω ε, ποιος είναι ο τρόπος που σκέφτεστε, πώς ε, τα προσεγγίζετε όλα αυτά και ίσως μπορεί να μας φωτίσει αυτό για τις διάφορες πτυχές ενός ενδιαφερομένου ή υποψηφίου για κάποια θέση. Και τέλος, ένα ερώτημα προς την κυρία Ανσόν. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι οι μελέτες σας δεν δείχνουν ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην επίδοση των επιχειρήσεων η ύπαρξη περισσότερων γυναικών. Αυτό το εξετάζεται από μικροοικονομική σκοπιά Δηλαδή, εξετάζετε τις εταιρείες μεμονωμένα σε επίπεδο μικροοικονομίας ή εξετάζετε και την μακροοικονομία. Από ό,τι καταλαβαίνω, η συντάκτες ε, ε, της μελέτες, της μελέτης από κοινού είναι και οι επίτροποι που έχουν οικονομικά χαρτοφυλάκια και άρα λαμβάνουν υπόψη τους και τη δημογραφική κατάσταση και εξετάζουν και το δυναμικό ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όλα αυτά φαίνεται να έχουν επηρεάσει αυτούς που συνέταξαν από κοινού τη μελέτη αυτή και θα ήθελα τη δική σας άποψη από αυτού. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τόμσον παρακαλώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Τις άκουσα προσεκτικά και νομίζω ότι οι ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις μπορούν να συναχθούν. Πρώτον προς την καθηγήτρια κυρία Γκόμες Άνσον. Είναι πολύ ενδιαφέρον, το είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, το παρατήρησε, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι είπατε ότι δεν υπάρχει διαφορά στις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Εγώ να σας πω ότι είστε σε επαφή μαζί μου ένα δανέζικο ραδιοφωνικό κανάλι, διότι ε, μας παρακολουθούν και ακούν τις δημόσιες συνεδριάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχα πει εγώ ότι με γυναίκες στις επιχειρήσεις έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό ε, δεν μπορούσε να αποδεχθεί. Όμως γυναίκες σε εκτελεστικές θέσεις έχει φανεί ότι έχουν μεγαλύτερες επιδόσεις στην οικονομία. Και σε αυτό το πλαίσιο ε, σκέφτομαι και το εξής και βλέπω ότι ασχολείστε με τα χρηματοπιστωτικά. 5% είναι οι γυναίκες παρούσες ε, δεν ξέρουμε αν ήταν 50%, 50 των επιτελικών θέσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αν καλύπτε το από γυναίκε, μήπω θα είχαμε αποφύγει τουλάχιστον το ίμιση αυτή τη κρίση που μα μαστίζει. Θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια που έχουν επιτελικές θέσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα εν γέννη. Και εγώ έχω μια ερώτηση να θέσω προς την κυρία Σίλβια Χόκροφτ. Έχω βαρεθεί να ακούω ε, για τις γυναίκες και την ε, οικογένεια. Εγώ 20% ε, των παιδιών στην Δανία είναι παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες, 75% όχι. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να τα λέμε αυτά. Εγώ για να δουλέψω άφησα τα παιδιά μου στην ηλικία των 43 ετών. Οι γυναίκες 45 με ταξί 65 μπορούν κάλλιστα να μην έχουν ε, παιδιά και να είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων. Ε, αυτά είναι πράγματι που ισχύει. Επίσης στην Ισπανία και στην Ιταλία τους ή άλλως δεν γεννάνε ε, και άρα δεν αφιερώνουν τη ζωή τους στην οικογένεια. Είναι ένα πλαστό επιχείρημα αυτό. Με έχει κουράσει ότι ε, οι γυναίκε ασχολούνται με την οικογένεια από την μέρα που γεννιούνται μέχρι τη μέρα που πεθαίνουν. Πρέπει να το αφήσουμε κατά μέρο αυτό το επιχείρημα γιατί δεν ισχύει. Και πρέπει να σα πω ότι ακόμα και τα κορίτσια παίρνουν μικρότερο χαρτζιλίκι από ότι τα αγόρια και βοηθούν τη μητέρα του στι δουλειέ του παιδιού περισσότερο από, τα, από ότι τα αγόρια. Το έχουν συνηθίσει δηλαδή. Και τελικά να σας πω ότι δεν συμφωνώ και με την Επιτροπή ως προς το 10%. Νομίζω ότι η βιομηχανία το έχει αυτό ε, εισαγάγει και δεν ισχύει. Θα πρέπει να έχουν γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια Ακόμα και στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό σύλλογο των Vikings στην Νορβηγία, το 40% στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ήταν γυναίκες. Γιατί, γιατί η επιχείρηση ήταν εισηγμένη, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα δηλαδή στην Νορβηγία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι κανόνες είναι ίδιοι εκεί που υπάρχουν λιγότεροι άνδρες. Όταν ένας ε- άνδρας μπαίνει σε μια επιχείρηση έχει ειδική αξία, π.χ. εκλέγεται πρόεδρο αμέσω. Το ίδιο ισχύει και στους νοσηλευτές, στο νοσηλευτικό προσωπικό. 2% είναι οι άνδρες νοσηλευτές έναντι των γυναικών νοσηλευτριών και όλοι οι επικεφαλείς εκεί είναι άνδρες. Φαίνεται ως να υπάρχει υψηλότερη ε, αξία όταν ένας άνδρας μπαίνει σε γυναικεία νερά. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει. Όταν μια γυναίκα μπαίνει σε ανδροκρατούμενα νερά, έχει μικρότερη αξία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει η γερμανική ε, βιομηχανία χάλιβα. Και όταν μιλούμε για την ενσωμάτωση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, εννοούμε και αυτού σε αυτή την ε, κρατεά βιομηχανία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιτ παρακαλώ. Κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί επιστημονικός και είναι απαραίτητο να μοιραζόμαστε την ευθύνη των παιδιών. Αυτό είναι πράγματι ουσιαστικό. Ε, και γι' αυτό το ανέφερα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Ίσως σας έχει κουράσει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Και πολλές επιστημονικές μελέτες το έχουν καταδείξει ότι η σταδιοδρομία είναι κάτι που μας απομακρύνει. Είναι μιλητή από το μικρόφωνο. Καλό είναι να ε, μιλήσει πιο κοντά στο μικρόφωνο. Παράκληση των διερμηνέων. Ε, νομίζω ότι έχει προστιθέμενη αξία να έχουμε περισσότερες γυναίκες ή ένα πολυλειτουργικό, εν πάση περιπτώσει, διοικητικό συμβούλιο, γιατί ενισχύει την ε, ανάπτυξη και την ύπαρξη πολλών οπτικών στη συζήτηση. Συμφωνώ. Όμως, σε μια ανταγωνιστική Ευρώπη χρειαζόμαστε νομοθεσία. Οι εταιρείε στη Φιλανδία και στη Σουηδία έχουν 35% γυναίκες και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία υπάρχει 2 ή 3%. Δεν είναι αντιγωνιστικό πλεονέκτημα να πούμε επενδύστε σε αυτές οι επιχειρήσει γιατί τα κάνουν καλύτερα και έχουν καλύτερε επιδόσεις. Θα πρέπει να εξισορροπηθεί η διαδικασία. Εγώ π.χ. είμαι επενδυτής. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το διοκτησιακό καθεστώς της επιχειρήσης. Συμφωνώ πολύ με αυτό που λέτε, όμως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σε ορισμένες χώρες είναι εθελούσιο το μοντέλο, και τα κάνουν τόσο καλά και έχουν τόσο καλές επιδόσεις όσο οι άλλες που έχουν υποχρεωτικό σύστημα. Δηλαδή ε, το ερώτημα μπορούν, μπορεί να απαντηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και η κυρία Κράτσα, τελευταία ομιλήτρια. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τις εμπειρογνώμονες ε, για, την πολύ, για τις πολύ ε, σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσαν και τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη για την αποτελέσματα ερευνών. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις που έχουν σχέση με την, όχι με την ευρύτερη προσέγγιση του θέματος ισότητος που θέλει πολλές ώρες και χρόνο να συζητηθεί αλλά που έχουν σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας. Πρώτον, εάν ε, μπορείτε να μας πείτε από τις μελέτες που έχετε κάνει σε διάφορες περιπτώσεις χωρών που ετοιμάζονται να εφαρμόσουν την οδηγία, ε, ε, μια νομοθετική προσέγγιση ή την έχουν ήδη εφαρμόσει, που έγκυται οι δυσκολίες η προετοιμασία των επιχειρήσεων τόσο στην κουλτούρα, τόσο στο μηχανισμό, τόσο στην εναλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για να μπορούν να εντάξουν γυναίκες μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια, πότε κάνουν εκλογές, πώς προετοιμάζονται για αυτές τις εκλογές των νέων μελών. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Και δεύτερον, ήθελα να σας ρωτήσω τα ανεξάρτητα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων. Από την εμπειρία σας είναι καλύτερο να προέρχονται από την επιχείρηση την ίδια, τουλάχιστον ένα ποσοστό, ή να είναι εντελώς ανεξάρτητα μέλη από την επιχείρηση. Αυτό αφορά άντρες και γυναίκες, αλλά μια και προβλέπουμε αλλαγές στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, ας δούμε και την προέλευση αυτών των, μελών, των νέων μελών που θα μπουν στα διοικητικά συμβούλια. Ευχαριστώ. Thanks Σας ευχαριστώ και θα δώσω τώρα το λόγο ε, στους ε, εισηγητές να απαντήσουν, στις εισηγήτριες, ε, να απαντήσουν σύντομα στις ερωτήσεις. Θα εκτιμήσω ιδιαίτερα την συντομία σας. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω με τις δύο ερωτήσεις. Ε, χαίρομαι κύριε Σμιτ που σας άρεσε το, η ομιλία μου, αλλά δεν ε, έχει πάντα δίκιο η αγορά. Η αγορά δεν βρίσκει πάντοτε τη σωστή λύση. Γι' αυτό πολλές φορές οι εταιρείες χρειάζονται ενθάρρυνση για να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, και χρειάζεται βεβαίως και ενθάρρυση να μπουν περισσότερες γυναίκες στην ιατρική και σε άλλα επαγγέλματα. Ορισμένα μοντέλα έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά, ε, ορισμένα όχι. Η εθελοντική δραστηριότητα εισήχθη επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ποσοστώσεις. Ε, αν οι δράσεις αυτές οι εθελοντικές είχαν ανελφθεί νωρίτερα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά την προετοιμασία των επιχειρήσεων ακριβώς, ε, εν ώψη της νομοθεσίας, ε, των υποχρεώσεων, των ποσοστώσεων και νέων στόχων, οι επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια. Ορισμένες επιχειρήσεις, ορισμένες εταιρείες χρειάζονται και επιμόρφωση το, η Ένωση Εργοδοτών ε, Επιχειρήσεων ε, στον Καναδά οργάνωσε τέτοια σεμινάρια, οργάνωσε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη θέση των επιχειρήσεων στον 21ο αιώνα για να ξεπεραστούν οι συνήθειες και τα παλιά μοντέλα προσλήψεων. Υπάρχει λοιπόν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να γίνεται σωστή αναζήτηση, ανοιχτή προβολή, ανοιχτή διαφήμιση της θέσης, σωστές ενέργειες και να εξετάζεται πάντοτε η συνολική ανάγκη του, του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι χρειάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Ας πούμε χρειάζεται ένα δικηγόρο, ένα νομικό σύμβουλο, ίσως όχι τρεις. Όσον αφορά τώρα την ανεξαρτησία, σε, πρέπει να γίνει η πρόσληψη, η κάλυψη της θέσεως εσωτερικά ή απ' έξω, δεν είμαι ειδική. Στο Ενωμένο Βασίλειο, εκεί έχω και την εμπειρία μου, οι περισσότεροι, τα περισσότερα ανεξάρτητα μέλη προέρχονται εκτός της ε, εταιρεία. Δεν αποκλείεται όμως και η άλλη επιλογή ε, το, η εκτελεστική ομάδα πρέπει να εξετάσει ισόρροπα τις υποψηφιότητες, αλλά εγώ πιστεύω ότι το μη εκτελεστικό μέλος, το ανεξάρτητο, όταν προέρχεται απ' έξω, παίζει ένα πολύ παραγωγικό ρόλο. Η κυρία Ανσόν, όσον αφορά την ε, μελέτη περιπτώσεως των επιχειρήσεων ε, δεν βασίζεται από δική μου μελέτη, αλλά από συμπεράσματα μελετών που ερεύνησα, που προϋπήρχαν και οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι ορισμένοι διαπιστώνουν μια θετική σχέση, ορισμένοι μια αρνητική σχέση και ορισμένη μια σχέση η οποία δεν, είναι, δεν έχει καμία σημασία, είναι ουδιαίτερη. Οι μελέτες που έγιναν στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας βρήκαν μια θετική σχέση μεταξύ απόδειξη, ε, μεταξύ των φίλων απόδοσης των φύλων ε, ε, γυναικών ανδρών. Υπάρχει λοιπόν ένα συσχετισμό στην απόδοση μεταξύ των φύλων. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι η διαφορά στο φύλο ε, βελτιώνει τις αποδόσεις ή ότι η διάκριση του φύλου δεν βελτιώνει την απόδοση. Εμείς ε, αυτό που θέλουμε είναι να αυξήσουμε τις θέσεις των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ε, βασιζόμενη σε μια ουδέτερη σχέση ε, μεταξύ συμμετοχής και απόδοσης. Γιατί θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε τις γυναίκες, διότι από τις μελέτες που έχουν προκύψει την τελευταία δεκαετία με βελτιωμένα στοιχεία, με βελτιωμένα δεδομένα ε, μεταξύ των 500 εταιριών του Forbes, ε, σκανδιναβικών εταιριών, δείχνουν ότι υπό μία χρονική περίοδο βελτιώνεται η απόδοση όταν συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες. Έχουμε λοιπόν τώρα αυτές τις επίκαιρα, τα επίκαιρα στοιχεία. Πώς βελτιώνεται λοιπόν η απόδοση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία έρευνα της αγοράς, αλλά τα αποτελέσματα διαφέρουν. Τα αποτελέσματα ε, κυμαίνονται. Δεν είναι πάντα τα ίδια όταν κάνουμε μελέτη αγοράς ή μελέτη αποδόσεων μιας επιχείρησης οι, γυναίκες πιστεύω πρέπει να συμμετέχουν στη δεξαμενή εργασία δεδομένου ότι έχουν πάρα πολλά ταλέντα αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η θεωρία του ταλέντου φτάνει επαρκεί για να δικαιολογήσουμε την περαιτέρω συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια. Χρειάζονται και άλλα στοιχεία. Τώρα, γιατί δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε γυναίκες μεταξύ 45 ας πούμε και 60 και το θέμα της οικογένειας των παιδιών. Εμείς θέλουμε να προσλαμβάνονται γυναίκες και άντρες με επαγγελματική εμπειρία. Το, το, η ύπαρξη των παιδιών ε, δεν είναι το μόνο στοιχείο, μπορεί να έχετε και ηλικιωμένους γονείς τους οποίους να πρέπει να φροντίσετε στο σπίτι και άλλα προσκόμματα που κάπως περιορίζουν την προσπάθεια στην καριέρα. Υπάρχουν λοιπόν γυναίκες που όταν τελειώνουν το MBA τους προσλαμβάνονται παρόλο που άντρες έχουν το ίδιο MBA σε χαμηλότερες θέσεις. Εντάξει, ίδιο πτυχίο, business administration αλλά χαμηλότερη θέση και εν συνεχεία μπαίνουν στην επιχείρηση, οι άντρες καρφαλώνουν γρηγορότερα και φτάνουν στις υψηλότερες θέσεις. Αν δεν λοιπόν τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, ε, και τους, ε, το διευθύνοντα σύμβουλο ε, και τους νομικούς συμβούλους και άλλους μπορεί πολλές φορές να λείπουν Α, ε, οι γυναίκες ως μη εκτελεστικές ε, διευθύντριες, διότι πολλά διοικητικά συμβούλια θέλουν να έχουν και εθνικούς ε, Υπηκόου και μόνο. Είναι και αυτό μία άλλη πτυχή. Και μαζί με την, προσε... την οτροπία. Και η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων Έχουμε εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά. Αυτό είναι μια σημαντική διάκριση. Όταν μιλάμε για μη εκτελεστικά μέλη, ε, είναι εκπρόσωποι μεγάλων, μεγαλομετόχων και ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δομή ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Στην Ευρώπη είναι αρκετά συγκεντρωτική. Έχουμε μεγάλα πακέτα ε, μετοχών και γι' αυτό ε, έχει σημασία να διαφοροποιούμε μεταξύ ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων μεγαλομετόχων. Να απαντήσω στις ερωτήσεις για τα ποσοστά των γυναικών. Αν ας πούμε κάνουμε μια έρευνα με 100 υποψήφιους, μόνο το 5% από τους 100 είναι γυναίκες. Δηλαδή 5% για αυτές τις εκτελεστικές θέσεις. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτό το 5% των γυναικών, οι περισσότερες λένε όχι δεν ενδιαφερόμαστε. Για τους λόγους που εξήγησα. Επομένως, οι δυνητικοί υποψήφοι ε, είναι πολύ λίγοι. Αυτό είναι μία από τις βασικές μου ε, συνεχεία. Σε ό,τι αφορά το, τις τεχνικές συνεντεύξεων ε, και το κατά πόσο ρωτάμε τα θέματα της οικογενειακής ζωής. Τα προβλήματα που έχουμε ως εταιρεία που ψάχνουμε τέτοια εκτελεστικά στελέχη είναι ότι περιοριζόμαστε από τις επιθυμίες του πελάτη. Ο πελάτης καθορίζει τους κανόνες για μας και μας πληρώνουν οι πελάτες. Επομένως θα πρέπει να τους δώσουμε ό,τι θέλουν. Αυτό είναι μία σταθερά, είναι δεδομένο. Αν Πάντα ρωτάμε, ας πούμε, τους υποψήφιους για την οικογενειακή τους κατάσταση, για το πλαίσιό τους, αν είναι παντρεμένοι, αν έχουν παιδιά, αν έχουν την κυθεμονία των παιδιών. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι άντρες, όταν είναι διευθυντές, αποκλείεται να πάνε να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο, να ασχοληθούν αν είναι άρρωστα. Και αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τότε ποτέ δεν πρόκειται να φτάσουν στη συνέντευξη ε, για ένα τέτοιο ρόλο, για μια τέτοια θέση. Οι γυναίκες με μικρά παιδιά θεωρούνται λιγότερο προσιλωμένες, ενώ οι άντρες με παιδιά θεωρείται ότι θα βρουν κάποιον που θα φροντίσει τα παιδιά τους, ότι έχουν μια λύση ήδη στο μανίκι. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν, δεν υπήρχαν νομίζω ερωτήσει προς εμένα. Τότε δεν χρειάζεται να πάρετε και το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Σας έδινα απλώ την ευκαιρία να απαντήσετε. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω μετά από αυτά που άκουσα. Μπορείτε να ξαναπάρτε το λόγο. Έχω, εγώ έχω μια ερώτηση προς εσάς κυρία Χόθορν όσον αφορά τα κριτήρια που είπατε, ευελιξία, ορθολογικό μυαλό, ε, κριτήρια, τα οποία είναι πολύ προσωπικά. Πώς, πώς χειρίζεστε αυτές τις απαιτήσεις, αυτές τις προδιογραφές, οι οποίες είναι υποκειμενικές, είναι στερεότυπες, ε, όταν λέμε ότι στη θέση αυτή πρέπει να είναι κάποιος ευέλικτος, πρέπει να είναι συνεργάσιμος, δημιουργείται μια συγκεκριμένη υποκειμενική εικόνα έναντι των αντικειμενικών προσόντων. Πώς το χειρίζεστε αυτό? Ευελιξία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των γυναικών. Το πρόβλημα με τις προϋποθέσεις, με τις απαιτήσει. είναι ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν είναι πολύ αντικειμενικές συχνά υποκρύπτονται άλλα πράγματα πίσω από αυτές. Ένας πελάτης, Φερρυπίν, θα πει ότι θέλει να προσλάβει κάποιον που είναι κάτω τα 100 εκεί, δεσμευμένος, προσιλωμένος στη δουλειά. Αν ας πούμε, πούμε, να αυτός έχει οικογένεια και είναι προσιλωμένος. Μπορεί να μην το προσλάβει. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε και τις προσωπικές μας αξίες, να τις περάσουμε. Αλλά δεν έχουμε εξουσία απέναντι στον πελάτη, ο οποίος θέλει να πάρει μια απόφαση με βάση τις δικές του προσωπικές προτιμήσεις, με βάση το ότι προτιμάει να προσλάβει. Μερικές φορές κρύβεται ο πελάτης πίσω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις που βάζει, ας πούμε, για το ποιο θα προσλάβει. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ και τις, τους ευρωβουλευτές που έκαναν ερωτήσεις. Ευχαριστώ τους ομιλητές που μας διέθεσαν το χρόνο τους και συνεισέφεραν στη συζήτηση. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, τις απαντήσεις σας. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο τμήμα του εργαστηρίου. Ε, αναλύουμε τις εθνικές καταστάσεις. Δηλαδή, ε, ποια είναι η νομοθεσία, ε, υπάρχουν ποσοστώσεις, ε, θελοντικά καθεστώτα. Πρώτος ομιλητής είναι εκπρόσωπος των συνδικάτων εταιριών που θα παρουσιάσει τη θέση μίας, ενός συνδικάτου και είναι η κυρία Κλάουντια Μένε από ETUC. Έχετε το λόγο. Δώστε μας ένα λεπτό να αλλάξουμε λίγο θέσεις. But maybe I can already use this time because it is, time is running short to present myself. As you said, I am member of... Ευχαριστώ. Είμαι... Είμαστε ένα εκλεγμένο σώμα. Ε, έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, 8 ατόμων, έχουμε 4 άντρες και 4 γυναίκες ε, στο δουσού μας. Ε, για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία μας ε, την ανώτατη επιτελική θέση την α, ε, κατέχει γυναίκα. Επομένως είμαστε συνεπείς, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Η ευθύνη μου είναι το εταιρικό δίκαιο, ε, θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών. Να ξεκινήσω ή να περιμένω για την ομιλία μου. Προχωρήστε. Θέλω να σας παρουσιάσω τη θέση της CTUC για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω καταρχάς να εδράσω τη θέση μου στην γενική μας άποψη για την πολιτική, να σχολιάσω την πρόταση που υπάρχει μπροστά μας και συνεχεία να μιλήσω για κάποια συγκεκριμένα θέματα και να σας ευχηστήσω την προσοχή αγαπητοί ευρωβουλευτές, στην ε, εκπροσώπηση που υπάρχει στα διοικητικά συμβούλια. Ε, δεν είναι προφανές ότι η ETUC έχει θέση για το ποια είναι τα εκτελεστικά στελέχη στα Δουσού. Βασίζουμε λοιπόν την ε, θέση μας στην πολιτική που είναι η καταπολέμηση της υποεκπροσώπησης, η καταπολέμηση της ανισότητας, ε, η καταπολέμηση των διακρίσεων αλλά υπάρχουν και διάφορα επιχειρήματα που, έχουμε, που έχουν ήδη αναπτυχθεί, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύουμε ότι έχουν δημιουργηθεί έτσι ένα σώμα επιχειρημάτων, μια επιχειρηματολογία υπέρ αυτής της ισότητας. Λοιπόν, υπάρχει μια επίσημη θέση της ETUC, είναι και δημόσια, υιοθετήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο αυτή η επίσημη θέση. Εν συνεχεία, ή μάλλον είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έγινε ε, από συμμετοχή γυναικών και, και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε γενικό επίπεδο η TUC και τελικά καταλήξαμε σε αυτή τη θέση τον Ιούνιο του 12. Στη θέση αυτή ε, επανυπεβεβαιώνουμε ότι οι εθελοντικές προσεγγίσεις δεν αποδείχτηκαν επιτυχείς, αυτό ακούστηκε ήδη. Πιστεύουμε ότι οι ποσοστώσεις δεν είναι αυτός σκοπός, ούτε ένα μόνιμο εργαλείο. Ο στόχος είναι να πετύχουμε την ισόρροπη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Οι ποσοστώσεις είναι ένα εργαλείο και όχι αυτός σκοπός, επαναλαμβάνουμε. Αυτός ο ε, αυτή η ρήτρα κατάληξης το sunset clause που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα. Φυσικά, ε, με βάση την προθεσμία, ε, ο στόχος είναι πάρα πολύ φιλόδοξος για το 2018 για τις ε, δημόσιες εταιρείες και το 2028 για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να υιοθετήσουν τη θέση και συνεχεία να την εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι οι σαφείς στόχοι, οι προθεσμίες και οι κυρώσεις θα πρέπει να συνεπάρχουν. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα από όλα αυτά. Θα πρέπει να τα έχουμε όλα. Και τα τρία αυτά στοιχεία. Στόχοι, προθεσμίες και κυρώσεις μαζί. Επανέρχομαι στη δική μας αρχή, που είναι ενδιαφέρουσα ίσως, ότι και εμείς εσωτερικά Εφαρμόζουμε αυτή την αρχή, ότι κάθε φίλο θα πρέπει να εκπροσωπείται ανάμεσα στο 40 και 60% σε θέσει που λαμβάνονται αποφάσεις, επιτελικές θέσει. Και σα έδειξα το παράδειγμα του δικού μα Διοικητικού Συμβουλίου και τη γραμματεία μα Προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτή την ισορροπία σε όλα μα τα όργανα και εκπροσωπούμε πάνω από 60 εκατομμύρια εργαζόμενους από τον κόσμο, 42 εκατομμύρια είναι γυναίκες. Ε, προσπαθούμε να πετύχουμε τουλάχιστον το 40% λοιπόν στις, στα δικά μας όργανα. Η θέση μας πάει λίγο πιο μακριά από την πρόταση που υπάρχει μπροστά σας, γιατί είπαμε ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να αφορά και τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων και θα πρέπει να αφορά την πλειοψηφία των εταιριών. Απαντήσαμε επίσης ε, και συμμετείχαμε μάλλον στη διαβούλευση της Κομισιόν και στη διαβούλευση είπαμε ότι πιστεύουμε στην ανάγκη να καλύπτουμε από την πρόταση περισσότερες ε, επιχειρήσεις. Ή τις περισσότερες επιχειρήσεις. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Είπαμε επίσης την διαβούλευση ότι αυτή η πρόταση δεν μιλάει μόνο για ποσοστώσεις ή για δεσμευτικά εργαλεία, κάτι που τόνισε ο κύριος Τσομπάνου, αλλά η πρόταση αυτή μιλά για μια διαδικασία προκειμένου να υλοποιήσουμε το στόχο. Και το θέμα είναι να εφαρμόσουμε διαφανείς στόχους ε, στις διαδικασίες προσλήψεων. Αυτό είναι από τα βασικά μηνύματα που προέκυψε ε, όταν συζητήσαμε αυτή την πρόταση και στην Επιτροπή μας. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να ακολουθείται από την αρχή συμμόρφωσης ή απολογισμού από τον εταιρικό κόσμο. Και επίσης ε, θα πρέπει να ενταχθεί στο εταιρικό δίκαιο των κρατών μελών αυτή η πρόταση. Πιστεύουμε ότι οι κυρώσει ή τα κίνητρα είναι πιθανά. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να έχουμε και θετικά κίνητρα, ας πούμε, για εταιρείε που εφαρμόζουν α, στους κανόνες τους στοιχεία αυτής της πρότασης. Πάμε στο συγκεκριμένο θέμα της εκπροσώπησης ε, των εργαζομένων. Είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, ίσως δεν το γνωρίζετε όλοι, γιατί υπάρχουν διαφορετικές μορφές εταιριών στην Ευρώπη. Έχουμε καταρχάς ε, τη διαφορά ανάμεσα στις κρατικές, ε, ιδιωτικές, εισηγμένες ε, στο χρηματιστήριο, εταιρείε που έχουν ένα εκτελεστικό όργανο ή περισσότερα. Έχουμε τη διάκριση ανάμεσα σε εκτελεστικά στελέχη και μη εκτελεστικά στελέχη. Αυτό όχι μόνο στη Γερμανία, τη χώρα μου, αλλά πάνω από 12 χώρε. χώρες. Κυρίως στις, α, κρατικές εταιρείες έχουμε περισσότερη συμμετοχή των γυναικών Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το είδος της εταιρεία στην πρόταση. Και πρέπει να έχουμε δυνατότητες προσαρμογής της πρότασης ανάλογα με τις εθνικές παραδόσεις. Για την εκπροσώπηση των εργαζομένων υπάρχουν διάφορες ε, διαδικασίες, εκλογές. Ε, γενικά υπάρχει δημοκρατική εκλογή. Ε, δηλαδή δεν ε, υπάρχει κυνήγη κεφαλών. Ε, πρόκειται για άτομα που προέρχονται από την εταιρεία, τα διευθυντικά στελέχη δηλαδή συνήθω. Επίση, ε, αν δούμε μόνο την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, από άτομα από την εταιρεία, ε, εργαζόμενοι τη εταιρεία, ε, εκεί το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο από τη και φτάνει μάλιστα στο 30% χάρη σε αυτές τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες, τις εκλογές δηλαδή που προβλέπονται. Ένα άλλο πιο λεπτό σημείο. Ε, πρέπει να είστε σίγουροι ότι η άποψή μας ε, διαφέρει από ό,τι ακούσαμε μέχρι στιγμή. Αυτά που ακούσατε ε, είναι διαφορετικά γιατί εμείς ας πούμε εκπροσωπούμε τα συνδικάτα και δεν έχουμε την ίδια κατανάγκη άποψη με άλλους που προέρχονται από εταιρείε κτλ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το επίπεδο γνώσης της εταιρεία. Όταν επιλέγουμε τα άτομα που θα εκπροσωπήσουν μια εταιρεία στο εταιρικό συμβούλιο, πρέπει να δούμε τη γνώση τους λοιπόν και θα πρέπει να δούμε και τα συμφέροντα ας που εκπροσωπούνται. Το θέμα της ανεξαρτησίας είναι θέμα ανησυχίας σε ορισμένε χώρες. Υπάρχουν όμως σχετικές αποφάσεις. Το θέμα της ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να είναι γενικά πρόβλημα. Τέλος. Κάνω έκκληση στους ευρωβουλευτές να συνεργαστούμε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να σεβαστούμε τις ε, εκλογικές διαδικασίες με βάση τις εθνικές πρακτικές ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τη δυνατότητα να έχουμε συγκεκριμένα ε, έδρες και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης ε, τα προσόντα των ατόμων που συμμετέχουν στα αυτά τα διοικητικά συμβούλια. Σας ευχαριστούμε κυρία Μένε γιατί μας ε, δώσατε την οπτική γωνία των ε, συνδικάτων. Η επόμενη ομιλήτρια θα μας παρουσιάσει τη θέση των μεγαλύτερων γαλλικών επιχειρήσεων. Η χώρα αυτή έχει θεσπίσει νόμου ποσοστώσεις πρόσφατα. Θα μας μιλήσει η κυρία Οντίλ Ντεμπρός, Διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας της ΑΦΕΠ, της Γαλλικής Ένωσης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, δεν είμαι εξπέριστα. στα τεχνικά θέματα. Εκπροσωπώ την ΑΦΕΠ. Είναι μια ένωση η οποία αποτελείται από τις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Γαλλίας, η Γαλλική Ένωση Ιδιωτικών Μεγάλων Επιχειρήσεων και θα ήθελα να σας μιλήσω πρώτον για τις συστάσεις ε, του κώδικα ε, διοίκησης της ΑΦΕΠ και της ΜΕΝΤΕΦ που ασχολείται με το θέμα των ποσοστώσεων και θα σας μιλήσω επίσης και για το νόμο έχουμε και soft law και hard law για τις ποσοστώσεις. Έχουμε δηλαδή και νόμο αλλά και νομολογία δικαστηρίων και είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο 40% στις προθεσμίες που έχουν τεθεί. Η κατάσταση στη Γαλλία είναι αρκετά καλή. Και στο τέλος της παρέμβασής μου θα σας δώσω κάποια στοιχεία για την εκτίμηση που κάνουμε ως προς την πρόταση οδηγίας που έχει τεθεί επιτάπητος. Επομένως, ως προς τον κώδικα ΑΦΕΠ-ΜΕΝΤΕΦ προβλέπει ότι ο στόχος είναι σε κάθε συμβούλιο διοικητικό να φτάσουμε σε ποσοστό τουλάχιστον 20% γυναίκες το 2013 και τουλάχιστον 40% γυναίκες στο, το 2016. Τι περιλαμβάνεται στις ποσοστώσεις αυτές. Όλοι οι διοικητές, όλα τα μέλη εποπτείας όταν πρόκειται για... Ε, εταιρείε. Δηλαδή περιλαμβάνονται και οι εκπρόσωποι διαχειριστές των εταιριών. Τώρα, ως προς τους μισθωτούς, το σύστημα είναι πιο περίπλοκο. Έχουμε δύο κατηγορίες διοικητών που λαμβάνουν μισθό. Έχουμε μισθωτούς διοικητές που εκπροσωπούν τους μετόχους, ε, όσοι έχουν 3% του εταιρικού κεφαλαίου και έχουμε και διοικητικές θέσεις τις οποίες εκλέγουν οι μισθωτοί ποιος θα πάει, οι υπάλληλοι. Η πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνεται λοιπόν στον καθορισμό των ε, ε, ποσοστώσεων, η δεύτερη κατηγορία μάλλον, διότι εξελέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Όσοι εκλέγονται άμεσα από τους υπαλλήλους δεν μπαίνουν στις ποσοστώσεις. Γιατί, Γιατί εκλέγονται από λίστες, καταλόγους που καταρτίζουν τα συνδικάτα. Επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να παρέμβει στο διορισμό και έτσι δεν μπορεί να αποφασίσει εάν χρειάζεται άνδρα ή γυναίκα. Επομένως, είναι προτιμότερο η δεύτερη κατηγορία να βγει από το σύστημα γιατί αλλιώς δεν θα ήταν αυτό εύκολο να γίνει αντικείμενο διαχείρισης βασιζόμαστε ε, στην αρχή ε, συμμορφωθείτε ή εξηγήστε. Comply or explain. Ε, πέρα από τη σύσταση έχουμε και τον νόμο που υιοθετήθηκε τον ε, Ιανουάριο του 2011 και ο οποίος εμπνέεται ιδιαιτέρως από την σύστασή μας. Ο νομοθέτης εμπνεύτηκε δηλαδή πάρα πολύ από τη σύστασή μας και είναι καλό αυτό για τις εισηγμένες επιχειρήσεις με την ίδια ποσόστοση ένας, ένα πρώτο σκαλοπάτι του 20% και ένα δεύτερο το 40% θα πρέπει να φτάσουμε στο 40% γυναίκες το 2017. Ο νόμος δίνει άλλη μια χρονιά πέραν του 2016 που βρισκόταν στη σύστασή μας και θα αφορά επίσης και τις μη εισηγμένες όταν όμως είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Έχουν ε, πάνω από συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού και το ισολογισμός τους ε, και ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνά ένα συγκεκριμένο κατόφλι. Προβλέπουμε μια κάπως πιο μακριά Μικροχρόνια προθεσμία, λογικό είναι, το 2020 για τις μη εισηγμένες. Τώρα, αναφερόμαστε σε όλα τα μέλη του Δικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εποπτείας, εξαιρώντας τους ε, ηθήνοντες που εκλέγονται από το προσωπικό, διότι αυτό δεν θα ήταν λειτουργικό, όπως καταλαβαίνετε. Από τη στιγμή λοιπόν που θεσπίστηκε νόμος, προβλέπονται και κυρώσεις. Ή θα ακυρωθεί ο διορισμός όταν δεν γίνεται σεβαστό το κατόφλι του 40% ή θα ε, δεν θα πληρωθούν η αποζημίωση για την ε, παραμονή στην ημερήσια συνεδρίαση του Δικητικού Συμβουλίου και δεν θα θεωρείται τακτική η συνεδρίαση αυτή. Ε, άρα είναι μια συλλογική κύρωση που θα πλήξει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν δεν τηρηθούν οι ποσοστώσεις και ο νομοθέτης εν τη σοφία του λέει ότι η ακυρότητα, ε, ο χαρακτήρας άκυρος της ε, θέσης δεν θέτει εν αμφιβόλο την εγκυρότητα της συνεδρίασης της, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιλούμε για εισηγμένε επιχειρήσει. Αν θεωρηθεί η συζήτηση άκυρη, αυτό θα έχει εξαιρετικέ επιπτώσει για του μετόχου κτλ. Και, και δεν θα έπρεπε να γίνει. Βλέπετε την κατάσταση στη Γαλλία τώρα σε αυτή τη γραφική παράσταση. Είναι αρκετά καλή η κατάσταση πιστεύω και η εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση σημειώνεται και μάλιστα ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ε, για τις εταιρείες που είναι στις πρώτες 40 θέσεις ε, του χρηματιστηρίου των Παρισίων πιστεύουμε ότι φτάνουμε στο 25,2 το 2012. Δεν μπορώ να σας δώσω τα αποτελέσματα για τα 13, θα το ξέρουμε τον Ιούνιο αυτό. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να φτάσουμε στο 26% ή και στο 27%. Πιστεύω ότι η έκπληξη θα είναι πολύ ευχάριστη τον Ιούνιο ως προς το 2013. Βλέπετε ότι προχωρούμε και είμαστε πιο μπροστά από ό,τι επιτάσσει ο νόμος, διότι ο νόμος είπε να φτάσουμε στο 20% γυναίκες το 2014. Άρα έχουμε ήδη διανύσει ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι προβλέπει ο νόμος. Αυτά λοιπόν η κατάσταση είναι σχετικά καλή θα έλεγα στη Γαλλία. Περνάω τώρα ε, στην οδηγία, την οποία και θα ήθελα να σχολιάσω. Επί της αρχής, ναι, γιατί όχι. Ούτως ή άλλως εμείς στη Γαλλία έχουμε νόμο από τη στιγμή που θα υπάρξει οδηγία και που δεν θα αντίκειται στο γαλλικό νόμο, βεβαίως και την ε, ε, καλοδεχόμαστε. Σίγουρα πρέπει να αποφύγουμε ε, εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες κατακαιρματισμένες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, με διαφορετικές κυρώσεις, με διαφορετική ισχύ δεσμευτικότητα, διαφορετικό βαθμό δεσμευτικού χαρακτήρα από τη μία χώρα στην άλλη. Βεβαίως και πρέπει να αποφύγουμε τους ποσοτικούς στόχους όταν μιλούμε για τους εκτελεστικούς ε, διευθυντές και εκτελεστικές διοικητικές θέσεις. Είναι θετική η προσέγγιση αυτή της οδηγίας, Ωστόσο, τα άρθρα της μας δημιουργούν τεχνικό πρόβλημα και θα ήθελα να μπω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες και ελπίζω να έχετε το κουράγιο να ακολουθήσετε το συλλογισμό μου. Για παράδειγμα, στους ορισμούς λέγεται κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κυρίως ένας εκπρόσωπος των υπαλλήλων, των μισθωτών. Στη Γαλλία αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει ή τουλάχιστον δεν μπορεί να λειτουργήσει κάθε φορά. Είναι καλύτερο εκεί να ε, έχουν τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αποφασίσουν ε, για τους ε, πρακτικούς τρόπους με τους οποίου θα γίνεται η εκλογή αυτού του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σίγουρα στη Γερμανία εκλέγεται ακολουθώντας διαφορετικό τρόπο το αντίστοιχο μέλος του ΔΣ συγκριτικά με τη Γαλλία. Άλλωστε, είναι προφανές ότι ε, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί οι ποσοστώσει. Δεν μπορούμε να έχουμε νέο νομοσχέδιο στη Γαλλία για τα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν για του ορισμού. Τώρα, στο άρθρο 4. Ε, ρυθμίζονται ορισμένε διαδικασίε οι οποίε μα δημιουργούν προβλήματα. Για παράδειγμα, άρθρο 4, εδάφιο 4. Λέγεται ότι τα κράτη-μέλη μεριμνούν έτσι ώστε οι εταιρείε όταν ε, απορρίπτουν έναν υποψήφιο που θα πρέπει να του παρουσιάσουν τα κριτήρια επιλογής, να κάνουν σύγκριση μεταξύ των αξιολογήσεων και ε, να πούνε ποια ακριβώς ήταν, ποιο ακριβώς ήταν το σκεπτικό που έκανε τη ζυγαριά να κλείνει προς τον υποψήφιο του άλλου φίλου. Αν δούμε το λεξικό, υποψήφιος είναι αυτός ο οποίος κάνει μια θετική δράση. Λέει ότι θα ήθελε να πάρει τυχή θέση. Δεν υπάρχουν αυθόρμητες υποψηφιότητες. Υπάρχουν βεβαίως βιογραφικά που στέλνονται, αλλά δεν στέλνονται τώρα για θέσεις διοικητικού συμβουλίου. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Οι επιτροπές διορισμού είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τους υποψηφίους σε συνεργασία με τα γραφεία κυνηγών κεφαλών, οι οποίοι κυνηγοί κεφαλών θα ε, ψάξουν για υποψηφίους βάσει ε, του επιθούμητου προφίλ της επιχείρησης. Ε, το να γίνεται συγκριτική και αντικειμενική αξιολόγηση ε, είναι κάτι το εξαιρετικά δύνατο. Πάντοτε υπάρχει υποκειμενικότητα όταν επιλέγεται ένας υποψήφιος. Άλλωστε, μπορεί το Συμβούλιο να μην επιλέξει, να υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διοριστεί κάποιος μέλος. Στη Γαλλία, ορισμένοι μέτοχοι, εάν ε, διαθέτουν και κατέχουν συγκεκριμένο ποσοστό μετοχών, μπορούν να υποβάλουν σχέδιο στη Γενική Συνέλευση για να ζητήσουν το διορισμό του χ διευθυντικού ή διοικητικού κτλ. Άρα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτή την περίπτωση, αυτά που περιλαμβάνονται οδηγία. Από εκεί και πέρα, στο πέμπτο εδάφιο λέγεται ότι, αναφέρεται ότι όταν ένας υποψήφιος δεν γίνεται δεκτός, τότε η εταιρεία θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν ε, ε, παραβίασε ε, τον κανόνα αυτό της ισότιμης μεταχείρισης, εάν υπάρχει τέτοια υποψία. Δηλαδή, υπο τίθεται να αμφιβόλω η σοβαρότητα της στρατολόγησης και της πρόσληψης ε, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ε, ε, ουσιαστικά γίνεται νομικήστικο εγχείρημα ο διορισμός του υποψηφίου. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία πιο άκαμπτη και να επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις. Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη μεριμνούν ώστε οι εταιρείε προβαίνουν σε ατομική δέσμευση για ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις εκτελεστικές θέσεις, ότι ατομικά δηλαδή επιχειρήσεις θα δεσμευτούν ότι θα έχουν ίση εκπροσώπηση. Με πάση ειλικρίνεια σας λέω ότι στις γαλλικές εταιρείες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι και ο μόνος εκτελεστικός εν μέσω μη εκτελεστικών. Σε ένα γαλλικό διοικητικό συμβούλιο με έναν πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο δεν βλέπουμε πώς μπορεί αυτό να γίνει ε, με ατομική δέσμευση. Στο γερμανικό σύστημα που έχουμε διευθυντήριο, ναι, εκεί μπορεί να έχουμε ανάληψη ε, δέσμευσης ατομικά. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως είναι η εταιρική κουλτούρα το εσωτερικό της χώρας μου. Από εκεί και πέρα έχουμε και πρόβλημα με τις ό Αυτό το οποίο αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο, ότι μια εταιρεία η δεν πληρεί τις αυτά θα πρέπει να εξηγήσει το γιατί και να περιγράψει τα μέτρα που έχει υιοθετήσει. Φαίνεται να προσωμιάζει σε αυτό το σύστημα του συμμορφωθείτε ή εξηγηθείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε ποια σχέση έχει και πώς διαρθρώνεται η παράγραφος αυτή με ένα άλλο εδάφιο του άρθρου 6, το οποίο προβλέπει καθεστώς κυρώσεων. Ή θα συμμορφωθούμε και θα εξηγούμε, αν δεν συμμορφωθούμε, ή θα θα κυρώσεις. Δεν μπορεί να γίνονται και τα δύο. Να, μου λένε λοιπόν ότι πρέπει κάπου εδώ να ολοκληρώσω, γι' αυτό και θα ολοκληρώσω κάπου εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιάστηκα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσετε τις γαλλικές θέσεις όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και τις διάφορες ε, αντι, που υπάρχουν και τώρα προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη και δίνω το λόγο στην καθηγήτρια Σίλβια Βόλμπι η οποία είναι από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και θα μας μιλήσει για τα υπάρχοντα νομικά μέσα ε, σε, για τις ποσοστώσεις ε, φύλου ε, στα διοικητικά συμβούλια. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Η συμβολή μου αναφέρεται στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών και των προσπαθειών τους να επιτύχουν μία ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων. Υπάρχουν εθελοντικοί και νομοθετικοί μηχανισμοί και σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών μηχανισμών, δηλαδή του εθελοντικού και του νομικού οι νομικοί, οι νομοθετικοί μηχανισμοί διαφέρουν ε, όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τις κυρώσεις, ε, τις διατάξεις και θα σας παρουσιάσω μερικά από αυτά τα συστήματα. Καταρχάς οι θελοντικοί μηχανισμοί. Εκεί ε, απαιτείται ειδική εκπαίδευση, δίδονται βραβεία και διάφορες αμοιβέ από τις εταιρείε. Υπάρχουν τράπεζες δεδομένων, τράπεζες στοιχείων που έχουν όλα τα στοιχεία για τις γυναίκες αυτές που μπορούν να παρουσιάσουν ε, εθελοντικά δηλαδή να αναλάβουν τέτοιες θέσεις και υπάρχει και το θέμα της αυτορύθμισης. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τρόποι υποστήριξης ενός εθελοντικού μηχανισμού. Αλλά η υλοποίησή του είναι σημαντική και έχει μεγάλες, ε, ε καθυστερεί πολύ και έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Τώρα, τα νομικά μέσα, οι νομικοί μηχανισμοί έχουν επιτύχει ένα 40% εκπροσώπησης γυναικών, ε, ε, χρησιμοποιώντας ποσοστώσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις κλπ, όπως η Νορβηγία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εθελοντικοί μηχανισμοί είναι άχρηστοι. Η βέλτιστη πρακτική είναι να εφαρμόζουμε και τους δύο μηχανισμούς. Και πραγματικά χρησιμοποιηθεί και οι δύο μηχανισμοί από τις χώρες που έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Αλλά χωρίς ε, το νομοθετικό υπόβαθρο καμία χώρα δεν ε, θα μπορούσε να έχει πλησιάσει το 40%. Αρκετές χώρες εφαρμόζουν τώρα αυτές τις ποσοστώσεις. Εννέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένες άλλες χώρες του ΟΣΑ. Ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών μελών έχει υιοθετήσει ποσοστώσεις πρόσφατα και βλέπετε από τον κατάλογο αυτόν Τη Δανία που υιοθέτησε τα μέτρα αυτά νωρίς, μετά την Φιλανδία, την Ιρλανδία και πιο πρόσφατα μία σειρά κρατών που υιοθέτησαν ε, τα, τις ποσοστώσεις το 2010-2011. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία το 2011. Υπάρχει λοιπόν μια αυξητική στάση υιοθέτηση ποσοστώσεων και γίνεται τελικά η εφαρμογή των ποσοστώσεων μια πρότυπη ευρωπαϊκή μέθοδος. Όσον αφορά τώρα τις διαφορές που σημειώνονται ε, υπάρχουν μικρές εταιρείες, μεγαλύτερες εταιρείες. Οι μικρές συνήθως αποκλείονται από αυτές τις ποσοστώσεις, ε, οι μικρομεσές, οι μεγαλύτερες ενδιαφέρονται. Επίσης υπάρχουν διαφορές στην δομή ιδιοκτησίας. Υπάρχουν κρατικές επιχειρήσεις, δημόσιες, ε, όπου το ενδιαφέρον του δημοσίου είναι μεγάλο και πρώτα εφαρμόζονται οι ποσοστώσεις αυτές στις δημόσιες επιχειρήσεις Εν συνεχεία υπάρχουν οι επιχειρήσεις που είναι συγμένες στο χρηματιστήριο, ανώνυμες ε, εταιρείε ΑΕ και εν συνεχεία υπάρχουν και επιχειρήσεις που εξαιρούνται που συνήθως είναι οι πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Στόχος λοιπόν της εφαρμογής των ποσοστώσεων είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλες εταιρείες, αε εταιρείες και εταιρείες δημοσίου δικαίου, δημόσιες. Όσον αφορά τώρα τους στόχους και το ποσοστό που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φάσμα κυμαίνεται μεταξύ 30-40%. 40% ε, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει επιλεγεί. Το, η οροφή. Ορισμένες χώρες έχουν εισαγάγει την ποσοστώσεις βαθμιαία. Καταρχάς λοιπόν είχαν μια μικρή ποσόστοση, ένα μικρό αριθμό και μετά ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά 40% αρχίζει και γίνεται πλέον μια, ένα το τυπικό ποσοστό της, μέσα στην Ένωση. Επίσης υπάρχουν και διαφορές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Συνήθως τις εταιρείε <clears throat> δίνονται μερικά χρόνια περιθώριο για να εφαρμόσουν αυτή τις νομοθετικές ρυθμίσεις και να υιοθετήσουν και το πλαίσιο κυρώσεων. Η εφαρμογή, όπως σας είπα, γίνεται πολλές φορές σταδιακά. Καταρχάς εφαρμόζεται ένα, ένας χαμηλότερος στόχος, πρώτα οι δημόσιες επιχείρησεις, μετά οι ιδιωτικές. Και πολλές φορές μεγάλες επιχειρήσεις πριν ακολουθήσουν οι μικρότερες. Η τάση λοιπόν είναι να επικεντρώνουμε τους στόχους μας στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κυρώσεων οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται μέσω των νόμων. Υπάρχουν λοιπόν κυρώσεις για επιχειρήσεις που έχουν παραβιάσει, βγαίνουν από το Μητρό ας πούμε, διαγράφονται από το Μητρό των επιχειρήσεων, επίσης ακυρώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο, απαλλάσσεται των καθηκόντων του, όπως ακούσαμε και από τη Γαλλία. Επίσης μπορεί ορισμένα μέλη του ΔΣ να χάσουν τα προνόμια τους ή να ακολουθηθεί μια διαδικασία κυρώσεων όπως προειδοποιητική, ένα προειδοποιητικό μήνυμα, συνεχεία πρόστιμο, μια άλλη κύρωση είναι ότι η εταιρεία χάνει την προτεραιότητά της στον κατάλογο των ε, αναθέσεων από το δημόσιο, αναθέσεως έργων, εργολαβικές δηλαδή αναθέσεις. Υπάρχουν πολλές ε, διαφοροποίησεις ε, στις κυρώσεις, στη μορφή των κυρώσεων. Νομίζω η πιο σημαντική διαφοροποίηση είναι το νομικό, οι νομικές θεμελιώδεις αρχές και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ενσωματώνεται η υποχρεωτική συμμόρφωση. Το νομικό καθεστώς, δηλαδή όλο το σώμα του νόμου που χρησιμοποιείται διαφέρει. Οι κύλοι υπάρχουν διαφορετικές ε, αρχές δικαιοσύνης, θεμελιώδεις αρχές του δικαίου που εφαρμόζονται Μέχρι τώρα η συζήτηση έχει επικεντρωθεί σε δύο αρχές. Η πρώτη είναι η κατάλληλη μεταχείριση ε, των υψηλόβαθμων γυναικείων στελεχών. Θα πρέπει να, να έχουν ίση μεταχείριση, να επιλέγονται λόγω της αξίας τους, και να υπάρχει μια θετική δράση υπέρ των γυναικών όταν υπάρχουν οι ίδιες ε, προδιαγραφές και τα ίδια προσόντα, τα ίδια κριτήρια στην πρόσληψη. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς το θετικό στοιχείο της ισότιμης μεταχείρισης με ένα μικρό σπρόξιμο υπέρ του φύλου. Λιγάκι δηλαδή θετική δράση υπέρ του φύλου. Και το βάρος εδώ τίθεται στην ε, δίκαιη μεταχείριση των γυναικών που ε, είναι στελέχη του ΔΣ. Η δεύτερη αρχή λοιπόν όμως η οποία αναφέρεται συχνά είναι το όφελος της επιχείρησης. Είναι προς όφελος της επιχείρησης να ε, έχει μία σωστή διακυβέρνηση. Και όταν μιλάμε διακυβέρνηση εννοούμε να έχει μία ποικιλομορφία το Διοικητικό Συμβούλιο, να μην χαραμίζονται ε, οι γυναικές στελέχοι που θα χαθούν μέσα στην επιχείρηση αν δεν ε, ενθαρρυνθούν και να μπορέσουν να ενθαρρυνθούν έτσι ώστε να λειτουργούν με όλο τους, ε, το, δυναμικό, με το καλύτερό τους δυναμικό. Μία τρίτη βασική αρχή και ήδη ανέφερα ότι ορισμένες εταιρείες έχουν προνόμια. Μία εταιρεία, παραδείγματο χάρη, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένη ευθύνη και έχει καταχωρηθεί έτσι, σημαίνει ότι οι μέτοχοι θα μοιράζονται τα κέρδη όταν η επιχείρηση είναι κερδοφόρος, όταν όμως η επιχείρηση έχει ζημίες, οι μέτοχοι προστατεύονται και οι ζημίε μεταφέρονται στους πιστωτέ, στο ευρύ κοινό και στις άλλες μικρές επιχειρήσεις που χρεοκοπούν. Υπάρχει λοιπόν προνομιακή θέση των ΕΠΕ, γι' αυτό λέγονται και ΕΠΕ, εταιρείε Περιορισμένης ευθύνη. Έτσι λοιπόν θα μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει. Υπάρχει μία δημοκρατική αξίωση να μπορεί κανείς να έχει το λόγο να αποφασίζει δηλαδή για την διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών προς όφελος του κοινού. Το, το κοινό δεν θα ωφεληθεί εάν οι επιχειρήσεις αυτές χρεοκοπήσουν, διότι θα χρεωθεί το βάρος της χρεοκοπίας. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα δημόσιο συμφέρον για την βέλτιστη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Και στο εταιρικό δίκαιο υπάρχει παράδειγμα στο καταστατικό επιχειρήσεων παραδείγματο χάρη στον ε, ε, επιχειρησιακό νόμο του 2006 του Ηνωμένου Βασιλείου όπου το δημόσιο συμφέρον έχει ενσωματωθεί στην νομοθεσία και λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο κοινό όφελος του ευρύτερου περιβάλλοντος της επιχείρησης η επιχείρηση λοιπόν πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο κοινό συμφέρον. Έτσι ώστε επιβάλλεται στην επιχείρηση για να σεβαστεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, να έχει ε, χρηστή διοίκηση, χρηστό και βέλτιστο διοικητικό συμβούλιο και όλες αυτές και η διάσταση αυτή που συζητούμε ενσωματώνεται σε αυτή τη χρηστή διοίκηση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και τέλος θα έχουμε μία ολοκληρωμένη ιδέα στα κράτη-μέλη. Θα προχωρήσουμε με, την μελέτη περιπτώσεων, με τις μελέτες περιπτώσεων και η πρώτη μελέτη το περιπτώσεως είναι της ε, κυρίας Κάτια Λάγκεμπούχερ από την, το Πανεπιστήμιο Γκέτε της ε, Φραγκφούρτης και θα μας ε, μιλήσει για τη διάσταση του φύλου και την ισότητα του φύλου στα διοικητικά συμβούλια της Γερμανίας. Θα ήθελα να μιλήσω για το τι χρειαζόμαστε όταν ε, εξετάζουμε την νομοθεσία και να δούμε τα διάφορα στοιχεία για τις κυρώσεις και τα λοιπά, για το είδος της συνεργασίας ε, για το οποίο μιλούμε. Όλα αυτά τα εξετάζουμε στη Γερμανία και συζητώνται. Και ερχόμαστε σε επαφή με τις μεγάλες επιχειρήσεις και ε, υπάρχει πρόταση να συμπεριληφθούν και αυτοί που έχουν υποχρεωτική συμμετοχή των υπαλλήλων. Στη Γερμανία οι σημαίνες επιχειρήσεις είναι διτές. Έχουμε δύο δηλαδή, δηλαδή διοικητικά συμβούλια. Έχουμε το διευθυντικό και το εποπτικό. Και θα ήθελα να ε, πω το εξή. Ποιο θέτει την ποσόστοση, όχι απαραίτητα ο νομοθέτη. Έχουμε το flexi quota, μια ευελικτοποσόστοση. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει συνεργασία για την απόφαση του ύψου τη ποσόστοση. Και μετά έχουμε και εξαιρέσει. Να μην υποτιμούμε τη δύναμη των εξαιρέσεων. Στα νομοσχέδια που συζητώνται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία θα δείτε ότι μπορεί να συντεχθεί ένας πολύ αυστηρός κανόνας. Μετά να προβλέψουμε πάρα πολύ ευρείες εξαιρέσεις και τελικά να είναι το αποτέλεσμα διαφορετικό. Για τις κυρώσεις ακούσαμε άλλωστε με τις κυρώσεις επιβάλλεται ο νόμος. Θα έλεγα ότι η διαφάνεια είναι το βασικό για να έχουμε ποσόστοση ή οτιδήποτε που να έχει σχέση με την ποσόστοση. Δηλαδή πλήττει τη φήμη. Η διαφάνεια έχει νόημα μόνο όταν θεωρούμε ότι πράγματι θα πλήξει τις εταιρείες και τη φήμη τους να πούνε ότι ε, δεν προσλαμβάνουμε γυναίκες. Τώρα, το ανακλητό ημί των μελών του Συμβουλίου που διορίζονται χωρίς να εκπληρώνεται μία απέτηση ποσόστοσης. Εμείς έχουμε μελετήσει το γαλλικό κανόνα και το είπε και η κυρία Ντεμπρός, ότι η θέση ανακαλείται, αλλά δεν ανακαλείται ότι έχει πράξει το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από μόνο του είτε έναντι τρίτων ε, μερών. Εάν διοριστεί ένα διοικητικό συμβούλιο και πούμε μετά ότι επειδή δεν υπάρχουν αρκετέ γυναίκε, δεν είναι έγκυρε οι πράξει τι οποίε έχει προβεί μέχρι τώρα και μπορούν να ακυρωθούν, ή και στο γερμανικό σύστημα μάλιστα να επανεκλεγεί, τότε πώς, ε, τι θα κάνουμε εναντί των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με τρίτα μέρη. Αυτά τα μέτρα λοιπόν ακύρωσης ε, είναι προβληματικά στο γερμανικό δίκαιο. Και τέλος ο αντίκτυπος στην πληρωμή. Έχουμε διάφορες ε, κυρώσεις, τις εξετάζει η οδηγία. Δεν τα περιλαμβάνει αυτά η γερμανική νομοθεσία. ας δούμε κάποιες νομοθετικές προτάσεις στη Γερμανία. Έχουμε το κώδικα εταιρική διακυβέρνησης, το οποίο μοιάζει με αυτό που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, έχουμε ένα μηχανισμό της συμμόρφωσης και της επεξήγησης. Τι λέγεται δηλαδή, πιο ήπια τακτική έναντι των διοικητικών διευθυντικών συμβουλίων όταν διορίζονται άνθρωποι στις θέσεις εκεί καλό είναι όσοι διορίζουν να εξετάζουν την πολυχρωμία αν θέλετε την ποικιλομορφία και να ε, δώσουν προσοχή στο φύλλο, αλλά χωρίς να οφείλουν υποχρεωτικά να το τηρήσουν και να το λάβουν υπόψη. Δεν εμποδίζεται δηλαδή κάποιος, κάποια εταιρεία να λέει ότι το τηρεί και να μην το τηρεί τελικά. Όμως τα συμβούλια τα επόπτικα ε, λέγεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να μεριμνήσουμε καταλήλως για την ε, εκπροσώπηση των γυναικών. Ο μηχανισμός δηλαδή απαιτεί από τις επιχειρήσεις να δηλώσουν ότι ναι, το κοιτάξαμε, το εξετάσαμε και είδαμε ότι όντως την πληρούμε αυτή την προϋπόθεση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διατύπωση και είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι να αμφισβητείται. κατά πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα. Τα πράγματα μόνο με αυτή τη διάταξη της ε, εταιρική διακυβέρνησης. Εξού και δεν μας εκπλήσει το ότι κυκλοφορούν διάφορα νομοσχέδια από τα πολιτικά κόμματα και γίνεται μια έντονη συζήτηση στα διάφορα υπουργεία στην Γερμανία. Ένα υπουργείο πιέζει για απέτηση ποσόστοσης, αλλά η Άγγελα Μέρκελ αυτή τη στιγμή δεν στηρίζει τόσο την ποσότητα ποσόστοση όσο αυτό το οποίο νομίζουμε φλεξικότα, ευέλικτο ποσόστοση αν θέλετε. Δηλαδή η ίδια η εταιρεία να αποφασίσει για την ποσόστοσή της. Στην ε, βιομηχανία του Χάλιβα δεν είναι πολλές οι γυναίκες στο εργασιακό δυναμικό. Είναι πιο δύσκολο να προσελκύσουμε τις γυναίκες στη δική μας επιχείρηση, άρα να επιβάλλουμε στη δική μας επιχείρηση μια ποσόστοση 10% γυναίκες. Και π.χ. σε τέσσερα χρόνια. Προχωράει λοιπόν η εταιρεία, δημοσιεύει την ποσόστοση που έχει η ίδια αποφασίσει και θα δούμε μετά αν θα εκπληρώσουν, θα τα καταφέρουν αυτό, ναι ή όχι. Έτσι, έτσι είναι αυτή η πρόταση για την ευελικτό ποσόστοση. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν υποβάλει ένα νομοσχέδιο και ένα άλλο μαζί με τους πρασίνους και ε, ζητούν περισσότερες ποσοστώσεις. Το νομοσχέδιο των σοσιαλδημοκρατών θέλει να φτάσουμε σε ποσόστοση 40% ενδεχομένως και το συνδυαστικό νομοσχέδιο των δύο θέλει να φτάσουμε το 40% το 2023 και προβλέπονται διάφορες εξαιρέσεις για τις μικρές επιχειρήσεις και σχεδόν καθόλου κυρώσεις. Αυτά συζητώνται αυτή τη στιγμή στη χώρα μου να σας πω τώρα ποια είναι η θέση των πανεπιστημιακών. Οι περισσότεροι δεν εγκρίνουν την πολιτική, την υφέρπουσα, λέγοντας ότι επειδή θεωρούμε ότι οι περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια θα αυξήσουν την ε, αξία της μετοχής. Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά αρκετές μελέτες δείχνουν ότι τελικά αυτό δεν αποδεικνύεται, δεν ακλώνεται η απόδειξη. Και δεν το επιθυμούμε τουλάχιστον στο εταιρικό δίκαιο. Και λέγεται ότι δεν είναι και συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διότι ε, αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, λένε. Ενθαρρύνει διακρίσεις σε συγκεκριμένους τομείς, και δεν υπάρχει και βάση στις συνθήκες, νομική βάση. Επικρατεί δηλαδή η συμπερισχή αρχή της επικουρικότητας και αυτό το οποίο ε, τονίζει η Επιτροπή δεν έχει σχέση με την κατάσταση της απασχόλησης. Δηλαδή είναι πολύ προβληματική για τους Γερμανούς νομικούς η νομική βάση που διάλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ με αυτού σε μεγάλο βαθμό. Και επίσης είναι ασύμβατο με το συνταγματικό δίκαιο της Γερμανίας και πάρα πολλοί νομικοί ειδικοί για εταιρικού δικαίου και συνταγματολόγοι βεβαίως, τονίζουν ότι το Σύνταγμα προστατεύει τους μετόχους ως προς το περιουσιακό τους στοιχείο. Άρα προβάλλουν το εξής επιχείρημα. Είναι δικαίωμα ιδιοκτησιακό του μετόχου στόχου να εκλέξει τα μέλη που θέλει να εκλέξει στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, ε, εταιρεία στον οποίο τις μετοχές κατέχει. Κανείς ε, κανόνας δεν μπορεί να πει σε μένα ως μέτοχο ότι πρέπει να εκλέξω χι γυναίκες εάν δεν θέλω να το κάνω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ ως ομιλήτρια, αλλά το συνταγματικό δίκαιο και το εταιρικό δίκαιο και πάρα πολλοί νομικοί ειδικοί συνταγματολόγοι και εργατολόγοι ε, και ειδικοί εταιρικού, εταιρικής νομοθεσίας συγκλίνουν σε αυτό. Και έχουμε και μια απόφαση δικαστηρίου από τη δεκαετία του 70 που είπαν ότι ε, ε, είναι καλό το ότι επειδή επιβλήθηκε υποχρεωτικά εκπροσώπηση από τους υπαλλήλους, αυτό ίσως είναι ε, προηγούμενο δικαστικό για να ισχύσει το ίδιο και για τις ποσοστώσεις των γυναικών. Αλλά δεν είναι σαφές αυτό ακόμα. Οι λόγοι τώρα τους οποίους οι γυναίκες δεν προχωρούν ε, δεν έχουν να κάνουν με αυτά τα νομικά. Έχουν να κάνουν με τα παιδιά, με, τα, ε, με τους ρόλους πρότυπα που επικρατούν στην κοινωνία κτλ. Δεν μπορούμε να κρατούμε τις επιχειρήσεις σε ομοιρία προκειμένου να πετύχουν στόχους που είναι στόχοι της κοινωνίας και που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη και που δεν έχουν τόση σχέση με το σκοπό για τον οποίο ιδρύεται μια επιχείρηση. Λένε λοιπόν κάντε ό,τι χρειάζεται ε, αλλά μην μας αναγκάζετε να προσλαμβάνουμε ανθρώπους ενώ δεν τους θέλουμε. Γενικά η νομική στη Γερμανία είναι πολύ επιφυλακτική ως προς αυτό, αλλά και η κοινή γνώμη γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θα ακούσαμε την περίπτωση της Γερμανίας και θα πάμε στην περίπτωση τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα παρουσιαστεί η μελέτη αυτή από την Έλενα Ντόλντορ, που είναι λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Queen Mary και επιστημονικός συνεργάτης στη Σχολή Διοίκησης του Κράνφιλντ. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ελπίζω να στείλω και μία χτίδα φωτός με αυτή την περιπτωσιολογική μελέτη. Εμείς είχαμε μία εθελοντική προσέγγιση στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από μία δεκαετία και στην παρουσίαση αυτή θα κοιτάξω κάποιες από τις επιτυχίες που είχαμε στη χώρα μου και κάποιες από τις προκλήσεις που ακόμα αντιμετωπίζουμε με την προσέγγιση που έχουμε επιλέξει. Καταρχά, να σα θέσω το πλαίσιο. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ότι γενικά το Ηνωμένο είχαμε μάλλον ε, θελοντική και όχι υποχρεωτική προσέγγιση στην εταιρική διακυβέρνηση. Οι εταιρείε υποτίθεται ότι θα πρέπει να ε, συμμορφωθούν με ένα κώδικα διακυβέρνηση που τον θέτει το Συμβούλιο Οικονομικών Αναφορών, που είναι η ρυθμιστική αρχή. Ε, και υπάρχει αυτή η αρχή συμμορφώσου ή εξηγήσου. Ε, το 2010 αναθεωρήθηκε ο κώδικας αυτός και βασίστηκε σε προηγούμενες μεταρρυθμίσεις και σε προηγούμενες εκθέσεις που είχαμε για αυτά τα θέματα. Μεταξύ των αρχών ε, για την καλή διακυβέρνηση μιλήσαμε για την αρχή της ε, ποικιλομορφία πολλές φορές. Ο σημερινός κώδικας ζητάει από τις επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη την ποικιλομορφία αυτή όταν κάνουν τις προσλήψεις και τους διορισμούς. Αυτή όμως η διάταξη ήταν αρκετά γενικόλογη και δεν συνοδεύεται από κυρώσεις. Πέρα από το νοματίζω και στυλιτεύω που συχνά το κάνουμε στον Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουμε άλλους μηχανισμούς πραγματικά ελέγχου. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω ότι η παρακολούθηση ε, λαμβάνει χώρα από το 1999 όταν έγινε η πρώτη έκθεση το, τότε ε, και επομένως δίδεται μεγάλη σημασία στο δημοσιοβίο για το αν συμμορφώνται οι εταιρείε ή όχι ή όχι. Η πρόσφατη έκθεση Davis για τις γυναίκες της, ε, στα Δουσού από τον Λόρδο Davis ε, ήταν πολύ σημαντική. Ε, έγινε μία δημόσια έτσι, έρευνα για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Ε, τι είναι το διαφορετικό που φέρνει αυτή η έρευνα. Είναι ότι καταρχάς η στρατηγική ήταν, βασιζόταν στη συμμετοχή πολλών ενδιαφερόντων, πολλών φορέων, ε, πολλοί επενδυτές, ε, ε, επιχειρηματίε, ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονε, πολιτικοί συμμετείχαν. Αυτό ήταν μια μοναδική εμπειρία. Και ένας συναδελφό μου ήταν στην Διευθύνουσα Επιτροπή που ετοίμασε αυτή την έκθεση, Επομένω, είχαμε πολλέ απόψεις Η έκθεση δημοσιεύτηκε τελικά σε αρχές του 2011 και ενίσχυσε την ε, προσέγγιση την εθελοντική, αλλά ε, προσθέθηκαν πάρα πολλά στοιχεία ε, σε σχέση με το παρελθόν, πολλές λεπτομέρειες. Καταρχάς, οι εταιρείε υποθέτουν θα θέτουν, πρέπει να θέτουν στόχους αναφύλλο, θα πρέπει να μετράνε τα ποσοστά ανδρών και γυναικών από τις ε, κατώτατες θέσεις μέχρι τις ανώτατες. Επίσης θα πρέπει να λένε ότι έχουν πολιτική διαφοροποίηση, ε, δηλαδή ύπαρξη και ανδρών και γυναικών στο, στα διοικητικά συμβούλια και τι κάνουν γι' αυτό, πώς το επιτυγχάνουν, πώς επιτυγχάνουν τους στόχους ε, που θέτουν οι ίδιες οι εταιρείε. Επομένως αλλάζει ο διάλογος, υπάρχει περισσότερος διάλογος, περισσότερη έμφαση, περισσότερη πίεση από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε αυτή η έκθεση το 2011 και ο Λόρδος ο Ντέιβις ο ίδιος ε, συζήτησε πάρα πολύ με επιχειρηματίες, με εταιρείε, έγινε πραγματικά μια αλλαγή στον Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι άλλαξε ποιοτικά ο διάλογος στο δημόσιο βίο, αλλά άλλαξαν τελικά και τα νούμερα από το 1999 που αρχίσαμε να παρακολουθούμε. Ήμασταν στο 6% ε, αριθμό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και σήμερα ο αριθμός αυτός έχει φτάσει στο 15%. Δεν είναι το ιδανικό νούμερο, αλλά υπάρχει πρόοδος. Και τα τελευταία δύο χρόνια επιταχύνθηκε η πρόοδος αυτή. Δηλαδή, πολύ περισσότερες γυναίκες προσλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το τι συνέβαινε την περασμένη δεκαετία. Τώρα, σε, όπως σε πολλές χώρες, ε, Στι εκτελεστικέ διευθυντικές διαθυντικέ έχουμε πολύ λίγες γυναίκες, επίμονα επίμνα 6 ε, με 7% ε, στις 100 πρώτες εταιρείε εισηγμένε στο Φούτσι. Ε, στις μη εκτελεστικέ θέσει έχουμε περισσότερες γυναίκες, έχουμε 22,4% και βλέπετε ότι υπάρχει ενωδική τάση επιταχυνόμενης επιταχυνόμενη από το 2010 και μετά. Άλλα ενθαρρυντικά σημάδια είναι ότι περισσότεροι διορισμοί αφορούν γυναίκες, περισσότερες γυναίκες διορίζονται, 25% σε νέες θέσεις που πήγαν σε γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια πέρυσι, ενώ το 2010 ήταν 13% το αντίστοιχο ποσοστό. Έχουμε 11 εταιρείε που έχουν ε, όλους που, που όλους τα μέλη είναι άντρες ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχουμε πάνω και έχουμε πολλές εταιρείες, 39% που έχουν πάνω από μία γυναίκα στο δουσού. Ε, αυτά ήταν για τις εταιρείες ε, που ήταν στο Φούτζι 100. Τώρα έχουμε μικρό... σε μικρότερε εταιρείε που συμμετέχουν στο δίκτυο χρηματιστηρίου Φούτζι 250. Ε, εδώ έχουμε διαφορετική κατάσταση. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Το πόσε γυναίκε υπάρχουν στα διοικητικά συμβούλια, πόσοι νέοι διορισμοί αφορούν τι γυναίκε, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, πόσο διαφανεί είναι οι διαδικασίε, ε, ποιο είναι ο ρόλο των εταιριών που αναζητούν νέα στελέχη, των κυνηγών κεφαλών α πούμε. Ε, Σας είπα ότι τον Ιούνιο του 2011, Ιούλιο 2011, δημιουργήθηκε αυτός ο εθελοντικός κώδικας ε, δεοντολογίας, χάρη και στην ε, συμμετοχή αυτών των εταιριών κυνηγών κεφαλών. Ε, εκεί αναφέρονται οι καλές πρακτικές. Ε, συχνά κατηγορούσαμε τις εταιρείες ότι είναι αδιαφανείς, ότι ε, ας πούμε, προσλαμβάνουν μόνο αγόρια εντό αγωγικών. Στη μελέτη που κάναμε, τώρα προέκυψε ότι υπάρχει περισσότερη όρεξη για να προσληφθούν και οι γυναίκες, ε, υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, ε, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο τι υποψήφιους ψάχνουμε, αυτό ο θελοντικό κώδικας επίση διοντολογία θέτει και στόχους. 30% ε, γυναίκες ε, ε, στον κατάλογο που παρουσιάζονται στους πελάτες είναι έτσι μια ήπια προσέγγιση θα έλεγα αυτή. Και προσπαθούν οι εταιρείε που αναζητούν τα στελέχη να το εφαρμόσουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει τώρα προσπαθούν να διευρύνουν το, την ομάδα πιθανών υποψηφίων. Προσπαθούν να σκεφτούν πρωτοποριακά καινοτόμα, ε, ψάχνοντας τα στελέχη. Ψάχνουν τις γυναίκες που είναι επιχειρηματίες, ε, που παρέχουν ε, υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι εφαρεντικά. Όμως ε, κάποιες πρακτικές που αποκλείουν τις γυναίκες συνεχίζονται. Ε, ασαφή κριτήρια επιλογής, φερρυπίν. Παραδείγματο χάρη ρωτάμε πώ μπορείτε να είστε αντικειμενικοί όταν ε, προσλαμβάνετε κάτι, κάποιον, όταν κολλάτε σε κάποια στερεότυπα. Επίσης, μερικές φορές οι, οι εταιρείε δεν ε, δαπανούν το χρόνο, ας πούμε, για να ζητήσουν ε, τις πιθανές γυναίκες υποψηφίους. Μερικέ φορέ επίση ε, υπάρχει μια συνενοχή με του πελάτε. Ε, όταν παραδείγματο χάρη ο πελάτη, ε, μιλάει γενικά και αόριστα α πούμε. Δεν προσπαθούν να τον πείσουν, ε, δεν προσπαθούν με αντικειμενικότητα κτλ. Ε, μερικές φορές ε, υπάρχουν υποψήφοι ας πούμε ε, που έχουν δώσει 8 και 9 συνεντεύξεις ας πούμε για τέτοιες διευθυντικές θέσεις. Ε, ενώ μέσω όρος μπορεί να είναι 2 ξέρω εγώ. Υπάρχει δηλαδή μια, υπάρχουν σαφή κριτήρια. Εν πάση αυτή τη στιγμή αναθεωρούμε αυτόν τον ε, εθελοντικό κώδικα και τον κυκλοφούμε περισσότερο. Με όλη αυτή την προσπάθεια, πού κατευθυνόμαστε στο Ενωμένο Βασίλειο. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 2020, έτσι όπως πάμε, θα πρέπει να έχουμε περίπου 35% γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια σε εταιρείε ε, του δίκτυ Foods 100. Αυτό θα γίνει μόνο εφόσον προοδεύσουμε με το σημερινό ρυθμό. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός, θα πρέπει η εμπλοκή όλων των διαφερομένων να γίνει πραγματικότητα και θα πρέπει οι νέοι διορισμοί, οι νέες θέσεις που αδειάζουν ε, να πηγαίνουν σε γυναίκες με τον ίδιο ρυθμό, αν όχι με μεγαλύτερο. Φυσικά ε, δεν υπάρχει μια σαφή στρατηγική, τα νούμερα ακόμα είναι χαμηλά. Θα πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις μικρότερες εταιρείε. Ε, στο, που ανήκουν στο FUTS 250, όπου η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια είναι πολύ χαμηλότερη. Ε, γενικά μπορώ να πω ότι οι ποσοστώσει τι αντιλαμβάνει το κόσμο με πολύ αρνητικό τρόπο. Τι παίρνει πολύ άσχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι λέμε ότι η δική μας προσέγγιση είναι θελοντική, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι laissez-faire, ότι είναι απόλυτα χαλαρή, ότι αφήνουμε εντελώ εταιρείε να κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, κάνουμε μία προσπάθεια με συμμετοχή όλων των διαφερομένων. Και παρότι υπάρχει απόρριψη των ποσοστώσεων από του επιχειρηματίε, όμω η απειλή ότι θα επιβληθούν ποσοστώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν πολύ αποτελεσματική γιατί τουλάχιστον γίνεται συζήτηση στο ΕΒ Τουλάχιστον προς αυτή την, από αυτή την άποψη σα είμαστε ευγνώμονε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε λοιπόν την ε, άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου, του ενημερώσαμε, μας ενημερώσατε για το Ηνωμένο Βασίλειο και ο τελευταίος ε, ομιλητής, η τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Μπεάτα Αναγκή από το Κορβίνους, Πανεπιστήμιο Κορβίνους της Βουδαπέστης. Ευχαριστώ πρόεδρε, είναι πάντοτε πολύ σκληρό, είναι δύσκολο να είναι κανείς ο τελευταίος ομιλητής ή η τελευταία ομιλήτρια, όμως έχω καλυφθεί σε πάρα πολλά σημεία από τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Προέρχομαι από το Κορβίνους το Πανεπιστήμιο Κορδίνου της Βουδαπέστης και διδάσκω κοινωνιολογία. Θα σας πω λίγα λόγια για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Αυτό το θέμα της ε, διαχείρισης της διάστασης του φύλου δεν ανήκει στις προτεραιότητες ε, της ε, δημόσιας και κοινής γνώμης. Η χώρα έχει εκπληρώσει τις περισσότερες υποχρεώσεις της εσωτερικά και εξωτερικά. Έχουμε μια αρχή διαχείρισης της διάστασης του φύλου, παραδείγματος χάρη έχουμε δρεώσει πούμε μια υπηρεσία, αλλά αυτό είναι όλο. Η θεμελιώδης αρχή της εφαρμογής της διάστασης του φίλου δεν ανήκει στις προτεραιότητες της πολιτικής ζωής στην Ουγγαρία και οι ίσες ευκαιρίες ε, παρουσιάστηκαν περισσότερο μετά την ένταξή μας. Ε, παρουσιάστηκε μεν η θεωρία ότι θα πρέπει να υλοποιήσει η διάσταση του φύλου, όμως στην πραγματικότητα είδα μία υποχώρηση των δεδομένων ε, όσον αφορά την παρουσία γυναικών. Η κατάσταση λοιπόν ε, του ρόλου των γυναικών και των γυναικείων θέσεων ήταν πολύ καλύτερη στην Ουγγαρία πριν από 28, πριν από 20 χρόνια. Ε, γι' αυτό Λοιπόν, η κατάσταση είναι πάρα πολύ λυπηρή και στεναχωρία με ιδιαίτερα, διότι υπολοιπόμασα τόσο πολύ έναντι άλλων. Διαπιστώνουμε λοιπόν τώρα ότι η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη στο παρελθόν. Πριν από 20 χρόνια, όταν άλλαζε το σύστημά μας, πολύ περισσότερες γυναίκες δούλευαν στην Ουγγαρία από ό,τι δουλεύουν σήμερα. Ήταν λοιπόν πολύ ψηλότερο το ποσοστό εργασίας γυναικών στην Ουγγαρία. Έχει πέσει τώρα σημαντικά. Επίσης υπήρχαν ε, ε, όλο και μεγαλύτερος αριθμός γυναικών που ανέβαιναν στις διοικητικές θέσεις και στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό τελείωσε αυτή η ιστορία σήμερα, διότι τότε υποστήριζε το κοινωνικό κράτος τις γυναίκες. Υπήρχαν θαυμάσιες εγκαταστάσεις ε, για τη φροντίδα των παιδιών, είχαν υποστήριξη κατά τη διάρκεια ε, το, της ε, ε, εγκυμοσύνης και μετά ας πούμε και μεγάλη, πολύ μεγάλη βοήθεια στην οικογένεια δηλαδή και στην ανατροφή των παιδιών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες μπορούσαν να εργαστούν και έπρεπε και να εργαστούν και επίσης η κοινωνία αποδεχόταν το ρόλο της εργαζόμενης γυναίκας. Δηλαδή ήταν κοινωνικά αποδεκτός ο ρόλος της εργαζόμενης γυναίκας. Αυτό έχει αλλάξει τώρα πάρα πολύ. όμως, ε, να πούμε και τα αρνητικά στοιχεία του παρελθόντος, ο άντρας δεν έπαιζε κανένα ρόλο στην ανατροφή ή στην υποστήριξη της γυναίκας. Βλέπαμε λοιπόν ότι οι γυναίκες ε, είχαν καταλάβει πολλές ανώτερες διοικητικές θέσεις. Γιατί, ε, διότι είχαν γίνει μεγάλες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις ε, ε, οφειλόταν ακριβώς και η επιτυχία των γυναικών. Ε, υποστηρίζονταν, χρηματοδοτούνταν τα ακαδημαϊκά, τα πανεπιστήμια, ακαδημαϊκοί φορείς κλπ. Και έτσι οι γυναίκες μπόρεσαν να προχωρήσουν. Όλη αυτή η κρατική υποστήριξη ήταν πάρα πολύ σημαντική στο Ανατολικό Μπλοκ. Επίσης ήταν ε, δυνατόν να μάθουν ξένες γλώσσες. Μπορούσαν να μάθουν θαυμάσια αγγλικά και γερμανικά ε, και έτσι να αυξήσουν τις πιθανότητες ανόδου πολύ περισσότερο από τους άντρες. Ε, οι έρευνες που έκανα δείχνουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Οπότε πολυεθνικές διεθνείς εταιρείε όταν άρχισαν και έφταναν και εγκασίστανταν στο Ανατολικό Μπλοκ και στην Ουγγαρία ε, παρουσίασαν θαυμάσεις ευκαιρίες ε, απασχόλησης των γυναικών. Δεν, δεν λέω ότι ε, αμέσως οι γυναίκες γίνανε υψηλόβαθμα στελέχη και managers και, και λοιπά. Ήταν πάντοτε στη δεύτερη βασμίδα, στην κατώτερη βασμίδα, όμως ήταν, κατελάμβαναν σημαντικές θέσεις στον οικονομικό τομέα και έτσι μειωνόταν το χάσμα και οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Τώρα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει και τώρα βλέπουμε ότι στις ανώτερες θέσεις οι γυναίκες έχουν χάσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας και αυτό το οποίο βλέπετε στη διαφάνεια είναι η, η δομή πυραμιδοειδής δομή των γυναικών που έχουν τριτοβάσμια εκπαίδευση, πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ότι γενικά απασχολούνται σε χαμηλότερα ε, διοικητικά επίπεδα και λείπουν οι γυναίκες αυτές και από τα διοικητικά συμβούλια και δεν υπάρχει καμία σε, ως ε, πρόεδρος συμβουλίου. Ίσως λοιπόν να εκπλαγείτε με αυτό το ποσοστό του 40% σε διοικητικές θέσεις των γυναικών. Εγώ, εμένα του, με εξέπληξε 35% είναι στην Ουγγαρία Α, και αυτό δεν οφείλεται στο ότι περισσότερες ε, γυναίκες ε, ανέβηκαν, προήξησαν σε ανώτερες θέσεις, αλλά είναι επειδή υπάρχει τέτοια κρίση οικονομική, πολλοί άντρες εγκατέλειψαν, είτε χάσαν τη δουλειά τους. Γι' αυτό ανέβηκε το ποσοστό των γυναικών. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε στην Ουγγαρία, ειδικά στο top management, είναι μια πάρα πολύ ισχυρά δεσπόζουσα ανδρική παρουσία. Οι άντρες δεσπόζουν και κανένα στην πολιτική ζωή δεν πιστεύει, δεν ασπάζεται δηλαδή το αξίωμα ότι πρέπει να προχωρήσουν οι γυναίκες και η διάσταση του φίλου κλπ. Επίση δεν υπάρχει αξιοκρατία. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για αξιοκρατία και για ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτά τα, τα, πράγματα που συμβαίνουν στην ευρύτερη κοινο, κοινωνία. Ε, αυτή λοιπόν η δομή της πυραμίδας στις επιχειρήσεις στην Ουγγαρία, στο management, δείχνει ότι η εκπροσώπηση των γενικών είναι ένα έκτο, ένα έβδομο έναντι των ανδρών, δηλαδή έχει πλέον ε, λιμνάσει η πρόοδος των γυναικών και τίποτα δεν γίνεται. Έχω συλλέξει μερικά στοιχεία από το μη περιορισμένο χρηματιστήριο της Βουδαπέστης. Είναι μικρό το χρηματιστήριο μας. 40 ε, εταιρείε ήταν εισηγμένες φέτος σε δύο κατηγορίες μοιράζονται και τα μόνα στοιχεία που θέλω να αναφέρω είναι η διαφορά μεταξύ της κατηγορίας Α και της κατηγορίας Β των εταιριών. Η κατηγορία Α των εισηγμένων περιλαμβάνει τις πιο δυνατές και μεγάλες επιχειρήσεις ε, με μεγάλη ρευστότητα και υψηλότερα η κεφαλαιοποίηση. Οι εταιρείες οι γυναίκες λείπουν σχεδόν, δεν υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία α των μεγάλων επιχειρήσεων, ανύπαρκτες. Και ε, βλέπετε ότι ακόμα και οι συγμένες επιχειρήσεις δεν έχουν υιοθετήσει, δεν έχουν ασπαστεί τη διάσταση του φύλου και πολλές φορές, ε, παρόλο που είναι δέκα άνθρωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι όλο ε, Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση και οι έρευνες που έχουμε κάνει εξηγούν, δικαιολογούν αυτή την κατάσταση. Αυτή λοιπόν η κουλτούρα που υπάρχει ως προς τη διάσταση του φίλου Έχει σχέση με την γενική νοοτροπία, τα ίση τα, τις συνήθειες, τα ίση και τα έσημα και πολλές φορές από κοινωνιολογικής πλευράς διαπιστώνουμε ότι η ουγγρική κοινωνία είναι πάρα πολύ παραδοσιακή και ε, διαχωρίζει σαφώς τους ρόλους των ανδρών ε, και των γυναικών. Οι γυναίκες δεν ε, πολλές φορές δεν δεν θεωρούν υποχρεωτική την εργασία, η κοινωνία δεν θεωρεί υποχρεωτική την εργασία των γυναικών. Ε, από τις έρευνες λοιπόν που κάναμε διοργανώσαμε ιδιωτικές και δημόσιες συζητήσεις σε ε, συγκεκριμένες ομάδες και διαπιστώσαμε ότι και άντρες και γυναίκες αλλά κυρίως οι άντρες είναι εναντίον των ε, διοικητικών θέσεων, εναντίον των γυναικών σε διοικητικέ θέσεις, δηλαδή στο management υπάρχουν ισχυρά, ισχυρές προκαταλήψεις και θεωρούν ότι οι γυναίκες που, που θέλουν να αναλάβουν διοικητικές θέσεις έχουν ανθρωπερπή χαρακτηριστικά, είναι σκληρές, φιλόδοξες και ανίκανες. Ε, οι γυναίκες επικρίθηκαν κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αν έχουν ε, μικρά παιδιά δεν επιτρέπεται να πάνε να δουλέψουν ας πούμε μετά από έξι μήνες, ε, δεν, αυτό είναι κακό και δεύτερον όταν φτάνουν σε μια ψηλή διοικητική θέση επικρίνονται, κριτικάρονται δηλαδή έντονα. Η, η κυβέρνηση είναι ε, ε, πολύ έντονα κατά της ρύθμισης των ποσοστώσεων δεν έχει γίνει καμία συζήτηση δημόσια, καμία συζήτηση ε, στην κοινή γνώμη ή στους πολιτικούς κύκλους και αντί να μιλάμε για τη διάσταση του φύλου, στην Ουγγαρία μιλάνε για οικογένεια, για αναπαραγωγικότητα των γυναικών κλπ. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να, να μπει η συζήτηση του φύλου στη δημόσια γνώμη, στην κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε την ε, περιπτωσιολογική μελέτη της ε, Ουγγαρίας. Δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι πρόεδρος κανείς, γιατί χρειάζεται να κόβει τους ανθρώπους που μιλάνε ξαφνικά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για συζήτηση. Θα ζητήσω την κυρία Ρέγνε, την κυρία Κράτσα, αν θέλουν να πούν κάτι πολύ σύντομα, πριν κάνω κι εγώ μια πολύ σύντομη ε, συνόψη της συζήτησης. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Ήθελα να πω ότι ήταν πολύ πλούσια η, η ανταλλαγή των απόψεων σήμερα το απόγευμα. Μπορεί να μην μιλήσαμε εμείς πολύ, να μην κάναμε πολλές ερωτήσεις, αλλά ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα ενδιαφέροντα σε όλους τους τομείς και από τις εμπειρίες των χωρών και από τις, ε, τα ευρήματα ερευνών και σίγουρα θα είναι χρήσιμα στην εργασία που θα κάνουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ bin noch kürzer. Vielen Dank für die äh, wunderbaren Präsentation. Θα ήθελα εγώ να πω ότι εδώ γίνονται, έγινε, έγινε μια θαυμάσια συζήτηση, ακούστηκαν πάρα πολλές δράσεις και έχει η πολιτική πλευρά πολλή ε, δουλειά να, να κάνει. Σας ευχαριστώ. Ας μιλήσω κι εγώ στα Σουηδικά. Δύο λεφτά θα κάνω. Σας υπόσχομαι. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω. όπως και οι δύο εισηγήτριε. και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές αλλά και τη γραμματεία για τη θαυμάσια δουλειά επιμελητίας που έκανε που, διοργανώντας αυτή τη διάσκεψη, αυτό το σεμινάριο και σας ευχαριστώ για την υπομονή που δείξατε όλοι ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους όλους όσους μίλησαν και όλους, όλους άκουσαν οι ομιλητές ε, μας είπαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Ευχαριστώ τις εισηγήτριες που τους εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον της εργασίας. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θαυμάσιο και τέλος και σημαντικό ε, για τις ποσοστώσεις μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις φυσικά πολύ λογικό. Είναι και θέμα επικουρικότητας στο κάτω-κάτω. Θα ήταν ενδιαφέρον ίσως να ακούσουμε και κάποιον που είναι κατά των ποσοστώσεων. Μπορεί να μιλάει ας πούμε για προσόντα, για γνώσεις. Και άρα οι ποσοστώσεις είναι κάτι το αρνητικό. Εμείς όμως μιλάμε γενικά για ποσοστώσεις. Αν κάποιος ε, είναι κατά των ποσοστώσεων, τότε θα πρέπει να είναι κατά και του σημερινού συστήματος. Γιατί και το σημερινό σύστημα σε ποσοστώσει βασίζεται. Αλλά τι ποσοστώσει, υπέρ των ανδρών. Οι άνδρες διαδέχονται τους άνδρες. Η μία φουρνιά ανδρών διαδέχεται την επόμενη. Την προηγούμενη, συγγνώμη. Αν σπάσουμε αυτό το σύστημα, μπορεί να το αντικαταστήσουμε με ένα άλλο το οποίο είναι πιο δίκαιο και απέναντι στις γυναίκες, που δίνει ίσες ευκαιρίες. Και με αυτές τις σκέψεις και προβληματισμούς θα ήθελα να τελειώσω. Ζητώ συγγνώμη που μίλησα τελευταίος, ε, μίλησα τελευταίος, μίλησα τελευταίος και είμαι και άντρας. Ε. Σας ευχαριστώ όλοι, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Καλή επιστροφή.